friends. Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω θερμά στην σημερινή ημερίδα που έχουμε με το Eurofound. Ως πρώτη αντιπρόεδρος της ε, Επιτροπής Απασχόλησης, σας καλωσορίζω εδώ με μεγάλη χαρά. Από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε πολύ στενές σχέσεις μεταξύ μας διότι μας προσφέρεται τόσα πολλά στοιχεία, νούμερα, δεδομένα που μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε στο δικό μας πολιτικό έργο εδώ. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα που έχουμε σήμερα. Εννοείται ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρουμε τι συμβαίνει εκτός των τυχών αυτών, αλλά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι από εμά εκπλαγήκαμε από τα αποτελέσματα των εκλογών στις Ηνωμένε Πολιτείες και οι σκέψεις μας μετά από αυτά τα αποτελέσματα με νέο πρόεδρο που θα έχουμε στις Ηνωμένε Πολιτείε. μας οδηγούν σε συμπεράσματα ίσως όχι τόσο εντυπωσιακά, αλλά ενδιαφέροντα. Οι δημοκρατικοί θεσμοί πρέπει να αποδεικνύουν στους πολίτες με μετρήσιμους τρόπους ότι μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους μέσω της πολιτικής. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να το προσπαθήσουμε και αυτό ακριβώς θα κάνουμε εμείς σήμερα με την σημερινή μας ημερίδα και θα προσπαθήσουμε την ευχή αυτή να την κάνουμε πραγματικότητα και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Ότι θέλουμε δηλαδή να κάνουμε πράγματα υπέρ των εργαζομένων. Και έτσι πολύ χαίρομαι που βλέπω τόσο πολλούς ε, παρόντες εδώ που αποφασίσατε να αρχίσετε την μέρα σας μαζί μας και να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε μέχρι αργά σήμερα το απόγευμα. Ας αρχίσουμε όμως με μια εισαγωγή από τον διευθυντή της Eurofound που είναι ο Juan Menendez Valdés. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω εδώ όλους σας εκ μέρους της Eurofound. Είμαι ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που και ιδιαίτερα στη δικιά σας επιτροπή που αποφάσισε να οργανώσει αυτή την ημερίδα. Ευχαρίστως συμμετέχουμε. Χαιρετίζω τον Τόμας Χέντερ που δεν είναι βέβαια μαζί μας εδώ σήμερα αλλά σίγουρα θα ενημερωθεί για το έργο μας. θα έχουμε εδώ πέρα και τον κύριο Πυρίνσκι και άλλους από τα μέλη εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε λοιπόν τις ε, συνθήκες εργασίες, πώς ε, αλλάζουν στην Ευρώπη και αν αλλάζουν προς το καλύτερο. Και να δούμε τι θέλουμε να πετύχουμε για να έχουμε καλύτερη εργασία στην Ευρώπη. Όλα αυτά είναι ζητήματα που δεν είναι βέβαια καινούρια. Οι συνθήκες εργασίας από την αρχή του σχεδίου ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης άρχισαν να μας απασχολούν. Θα επαναλάβω αυτά που λέει το άρθρο 151 της συνθήκης για την βελτίωση συνθήκων ζωής, ότι αυτές συνδέονται με την απασχόληση. Και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας βέβαια αποτελούν το έμβλημα της Eurofound. Αυτό είναι ο στόχος μας. Αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Ακόμα λοιπόν και αν όλοι αυτοί οι στόχοι δεν είναι νέοι και πάντα τους είχαμε, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν και σήμερα. Καθ' άλλο. Σήμερα, αν λάβουμε υπόψη μας τις εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες, όλα αυτά αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία σήμερα. Ξέρουμε ότι έχουμε περάσει από την πιο βαθιά ευρωπαϊκή κρίση πρόσφατα που ξεκίνησε ως οικονομική κρίση, στη συνέχεια ως νομισματική και στη συνέχεια κοινωνική κρίση και κατέληξε σε χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς και απέναντι στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η απασχόληση είναι σημαντική και στην ε, μικρή αυτή ανάκαμψη που διαπιστώνουμε σήμερα, διαπιστώνουμε ότι και η απασχόληση βελτιώνεται, λίγο βέβαια, και όχι σε όλες τις χώρες μέλη. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολλές δυσκολίες εκεί. Έπειτα η ποιότητα ε, παίζει ρόλο στην απασχόληση. Χρειάζονται καλές συνθήκες εργασίας, γιατί έτσι συνάδουν με την καλή ποιότητα ζωής για τα εκατομμύρια τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Ενώ ανάποδα, αν δεν υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας, αυτές δεν μένουν στην δουλειά όταν γεννάμε σπίτι, όχι. Τις κουβαλάμε μαζί μας γιατί επηρεάζουν ολόκληρη τη ζωή μας. Συνεπώς, η ποιότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία στη δουλειά αν θέλουμε οι Ευρωπαίοι να εργάζονται περισσότερο. Και ξέρουμε ότι αυτό αποτελεί μια πρόκληση και μια δυσκολία για τις κοινωνίες όπως είναι οι ευρωπαϊκές που γερνάνε περισσότερο. Άρα πρέπει να τα καταφέρουμε περισσότερο, καλύτερα. Το καλό νέο είναι ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε στη ζυγαριά την ποιότητα της απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα καθόλου. Αυτά τα δύο μπορούν κάλλιστα να πάνε μαζί, γιατί μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους, που είναι το ανθρώπινο κεφάλαιό μας, ώστε αυτοί να προχωρήσουν σε καινοτομίες και σε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα. Το κακό όμως νέο είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, κοιτώντας την ποιότητα της απασχόλησης των Ευρωπαίων εργαζομένων, 20% περίπου από αυτούς λένε ότι έχουν απασχόληση που δεν θεωρείται ποιότητας. Και αυτό σημαίνει πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Όσοι δηλαδή είναι και κάτοικοι της δικιάς μου της χώρας της Ισπανίας, που είναι μια μεγάλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, εμείς στη Eurofound πρέπει να προσφέρουμε τα στοιχεία, τα δεδομένα, τη γνώση που χρειάζεται για την εκπόνηση καλύτερων πολιτικών και πολιτικών που θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και εργασίας. Η σημερινή διάσκεψη χρησιμεύει ακριβώς για να σας παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή, την ε, έκτη έρευνα για τις συνθήκες εργασίας και ζωής, που είναι μια από τις πιο σημαντικές πηγές δεδομένων που μας επιτρέπει να φέρουμε και σε πέρα στην εντολή μας που είναι να σας ενημερώσουμε για να αποφασίσετε πάνω σε καλύτερες πολιτικές. Πρέπει να καταλάβετε πρώτα απ' όλα την απασχόληση και την ποιότητά της στην Ευρώπη και όχι μόνο, και πέρα από την Ευρώπη. Ξέρω ότι την έκθεση αυτή τη χρησιμοποιεί η Επιτροπή σας, αλλά και όχι μόνο, και άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινωνική Εταίρη, χώρες μέλη αλλά και σε διεθνές επίπεδο αποτελεί μια πηγή που χρησιμοποιεί, το όσα, ε, που χρησιμοποιεί όσα. Προσφέρει στοιχεία τα οποία είναι πολύτιμα για πολλές πρωτοβουλίες που συζητάτε εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αλλού. Για παράδειγμα, το στρατηγικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ή η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή, ένα πακέτο συμφιλίωσης των δύο, που αποτελεί μέρος του πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα. Αρχίσαμε, όχι εγώ μάλλον, αρχίσανε, εγώ δεν ήμουν ακόμα εκεί, αρχίσανε πριν από 25 χρόνια στη Eurofound με την έρευνα αυτή. Και έχει αλλάξει βέβαια πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Αρχικά ε, πρόκειτο μόνο για κάτι σαν βαρόμετρο. Είχαμε 30 ερωτήσεις όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Το 2015 ήδη είχαμε πάνω από 100 ερωτήσεις που ταξινομήσαμε όσο γίνεται καλύτερα για να έχουμε μια έγκαιρη περιγραφή της πραγματικότητας στην εργασία και έτσι να έχουμε μια εικόνα τη ζωή στην εργασία από αυτούς που είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, αυτοί που εργάζονται κάθε μέρα, από τους εργαζόμενους δηλαδή. 54.000 συμμετείχαν, 45 λεπτά συνέντευξη για να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που αποτελούν πολύτιμες πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα την κατάσταση της εργασίας. Η συνολική εικόνα λοιπόν που παρουσιάζει η έκτη αυτή έκθεση δεν ε, δείχνει τίποτα δραστικές αλλαγές. Η συμμετοχή των γυναικών έχει αυξηθεί, έχει ε, μεγαλύτερη ηλικία κατά μέσο όρο το εργατικό δυναμικό. Ο μέσος όρος του εργαζόμενου Ευρωπαίου είναι με σύλικας, άντρες, με μόνιμη απασχόληση που εργάζεται σε τακτικές ώρες. Και όσον αφορά άλλες ηθικές εργασίες, είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά του, νιώθει στήριξη από τους ε, συναδέλφους του και από τους ανώτερους και μαθαίνει στη δουλειά του. Όμως, πολλοί από αυτούς λένε ότι δουλεύουν πολύ εντατικά ότι η ισότητα δεν τηρείται, ότι μερικές φορές υπάρχουν και κίνδυνοι για τη φυσική τους ακεραιότητα και πολλές φορές αντιμετωπίζουν δύσκολες κοινωνικές ε, συνθήκες, κοινωνικό περίγυρο. Κάτι το οποίο βέβαια επηρεάζει πολύ το θέμα της ικανοποίησης στην εργασία. Εμείς ε, βέβαια κοιτάμε τους μέσους όρους. Αυτό όμως κρύβει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των 35 χωρών στις οποίες κάναμε την έρευνά μας, τις διαφορές και μεταξύ χωρών αλλά και μεταξύ ατόμων και μεταξύ των δύο φύλων και μεταξύ των τομέων απασχόλησης, των ηλικιών κλπ. που είναι επίσης πολύ σημαντικά να λάβουμε υπόψη μας. Η έκτη αυτή έκθεση μας δείχνει ένα επίπεδο που είναι κατά πάσα πιθανότητα το υψηλότερο όσον αφορά τη διαφοροποίηση στον χώρο εργασίας. Ο κόσμος αλλάζει και ο κόσμος της εργασίας επίσης αλλάζει. Δεν γίνεται πιο απλός, αντίθετα γίνεται περισσότερο περίπλοκος. Θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Οι αυτοπασχολούμενοι. Πρόκειται για άτομα που μερικές φορές και είναι αρκετές αυτές, δεν ξέρουν ακριβώς ποιο είναι το καθεστώ τους. 13% αυτών των αυτοπασχολούμενων έχουν έναν απευθείας πελάτη, δεν μπορούν να προσλάβουν ή να απολύσουν κόσμο ή να πάρουν σημαντικές αποφάσεις. οικονομικά τελικά είναι εξαρτώμενοι. 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σημαντικό. Δεύτερο παράδειγμα. Ο χώρος απασχόλησης δεν είναι κάτι προφανές. 11% των εργαζόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν τις ε, τεχνολογίες πληροφορικής για να εργάζονται. Τουλάχιστον 3 τέταρτα του χρόνου τους κάθε μέρα ή πολλές φορές την εβδομάδα εργάζονται στο σπίτι τους, στο αυτοκίνητό τους, εκεί που είναι οι πελάτες τους, σε άλλους χώρους. Και οι συνθήκες εργασίας είναι βέβαια διαφορετικές από τις συνθήκες εργασίας όταν κάποιος κάθεται, όπως γινόταν παλιά, στο γραφείο του πάντα. Υπάρχει βέβαια κάποιο κέρδος, γιατί υπάρχει έτσι μεγαλύτερη ευελιξία. Από την άλλη μεριά όμως, η ισορροπία ανάμεσα στην ε, προσωπική ζωή και την εργασία δεν τηρείται πλέον. Και κάποια άλλα παράδειγματα θα μπορούσα να δώσω για να σας δείξω πόσο αλλάζει ο εργασιακός χώρος και κάτι το οποίο δεν φαίνεται από τα μεγάλα νούμερα. Όσοι παίρνουν τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εθνικές κυβερνήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι, οι διάφορες ε, οργανώσεις, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αλλαγές αυτές για να κατανοήσουν καλύτερα την ποιότητα της εργασίας και πώς ε, ζουν την εργασιακή τους εμπειρία οι πολίτες μας. Στη σημερινή διάσκεψη θα σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα μιας πρώτης συνολικής ανάλυσης της ε, έρευνάς μας αυτής. Πριν από μερικούς μήνες υπήρξαν τα αποτελέσματα, τώρα θα έχετε την ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών. Και επιπλέον, πέρα από τα στοιχεία δηλαδή και την ανάλυση, σας ζητήσαμε να συμμετέχετε στα πάνελς και να συζητήσετε μαζί μας για τα θέματα τα οποία θα καλύψουμε για να σκεφτούμε πολιτικές απαντήσεις στα διάφορα φαινόμενα. Θα αρχίσουμε με ένα πρώτο πάνελ, με μια πρώτη μάλλον παρουσίαση του κυρίου Τερών, α δεν είναι ακόμα εδώ, του, της κυρίας Ανιές Τυριών, η οποία θα παρουσιάσει τις διάφορες διαστάσεις που έχουν σημασία για την ποιότητα της απασχόλησης. Θα σας δείξει τι προφίλ έχει η Ευρώπη βάσει της ποιότητας εργασίας. Η ποιότητα εργασίας μπορεί κανείς να τη δει σαν μια εικόνα η οποία όμως δεν παρουσιάζει την εξέλιξη ενώ στη συνέχεια στο πάνελ θα συζητήσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν το εργασιακό περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ζωής μας, οι αλλαγές, η σταδιοδρομία κτλ. Και θα επικεντρωθούμε κυρίως στο θέμα της ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Σήμερα το απόγευμα θα επεκτεθούμε ακόμα περισσότερο και δεν θα περιοριστούμε στην Ευρώπη, αλλά θα πάμε πιο πέρα. Γιατί η ποιότητα της απασχόλησης φυσικά και έχει σημασία για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη, αλλά έχει σημασία και για τους εργαζόμενους παντού στον κόσμο. Σε μια παγκοσμιοποιημένη ανταγωνιστικότητα αυτό έχει σημασία. Δεν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο και μάλλον θα δούμε κατά πόσο οι συνθήκε εργασία, η ποιότητα εργασία παίζει ρόλο σε αυτήν την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε θα κοιτάξουμε εκτός από το τι κάνει η Ευρώπη, τι κάνουν και άλλοι εκτός Ευρώπης στον τομέα αυτό. Θα μιλήσουμε λοιπόν για όλες αυτές τις προκλήσεις πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε περισσότερο, περισσότερα χρόνια στην εργασία τους εργαζόμενους, πώς θα φροντίσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά κυρίως πώς η ανεργία και οι κακές συνθήκες εργασίες οδηγούν τους ανθρώπους να δείχνουν δυσπιστία και έτσι να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις, ε, στα δικά τους τα καθήκοντα τα εργασιακά, αλλά και πώς δυσκολεύεται η ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και εργασιακή ζωή. Ωραία. Τώρα, Ανιές, Ανιές, σε βλέπω, σου δίνω το λόγο για να παρουσιάσεις την ανάλυση και τα αποτελέσματα. Okay, I start again. Uh, Good morning, everybody. The question that Madam Chair asked us at the beginning is how can we improve um, people's life? Well, Λοιπόν, ένας από τους τρόπους βελτίωσης της ζωής μας είναι η ποιότητα της εργασίας. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος ε, για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ε, πολιτών. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη γιατί μπορώ να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της έκτης πανευρωπαϊκής έρευνας για τις συνθήκες εργασίας. Καλύπτουμε ε, την, ε, εκτός από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τις πέντε υποψήφιες, την Νορβηγία, την Ελβετία. Έχουμε παραπάνω από 43.000 συνεντεύξεις και ευχαριστώ την Ισπανία, το Βέλγιο, και την Σλοβενία που μας εμπιστεύτηκαν και που χρησιμοποιούν σε εθνικό επίπεδο τα αποτελέσματα της έρευνας. Πρόκειται για την μεγαλύτερη συγκριτικά έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για τεράστια πηγή πληροφοριών και είναι σημαντικό λοιπόν να εστιάσουμε σε αυτήν. Τεχνικά δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουν οι διαφάνειες. θα σας ε, δώσω μια απεικόνηση των συνθήκων εργασίας στην Ευρώπη ε, και σας λέω λοιπόν ότι για πέντε λόγους εμείς θέλουμε να εστιάσουμε στην ποιότητα των, της απασχόλησης. Πρώτον, τα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ε, έχουν ήδη σαν στόχο θέση τη βελτίωση της ζωής και των συνθήκων εργασίας. Δεύτερος λόγος είναι γιατί η ποιότητα της εργασίας συνδέεται με τον βαθμό ε, απασχόλησης και αυτό είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Η μακροβιότητα δηλαδή των θέσεων εργασίας είναι πολύ σημαντική. Τρίτος λόγος, μέχρι τώρα έχουμε λίγα στοιχεία, αλλά πάντως ε, γνωρίζουμε ότι σε επίπεδο, σε επίπεδο μικρής κλίμακας βελτιώνεται η υγεία εάν η ποιότητα εργασίας είναι καλή. Επόμενο στοιχείο είναι ότι η σωστή ποιότητα, η καλή ποιότητα απασχόλησης μπορεί να υποβοηθήσει άλλους στόχους στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, Πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε μελλοντικές εξελίξεις και μελλοντικές ε, αλλαγές. Πρέπει να το δούμε σαν ένα είδος φάρου ε, που μπορεί να μας ε, οδηγήσει σε ασφαλέστερους λιμένες στο μέλλον, να μας οδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε να μελετήσουμε το ε, θέμα της ποιότητας. Ε, τι προκύπτει από την έρευνα, ότι η ποιότητα της εργασίας ε, είναι πολυδιάστατη. Θα σας δείξω ότι δεν είναι αφηρημένη έννοια ή απλή λέξη η ποιότητα εργασίας. Ε, ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ε, σύμφωνα με το είδος της απασχόλησης, ε, με το φύλλο που διαφοροποιούν την ποιότητα. Δεν είναι καθόλου αφηρημένη έννοια. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουμε αναπτύξει κάποιους δείκτες και ευχαριστώ τον Φράνσις Γκριν και τον συνεργάτη του Τέρεκ Μουσταφά για την βοήθεια ε, κάθε διάσταση ε, υποστηρίζει ε, μια θετική εμπειρία της εργασιακής ζωής. Τρίτη ένδειξη είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε πολύ μεγάλη εξέλιξη και πρόοδο όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας. Έχουν υπάρξει βεβαίως πρόοδοι, αλλά ε, ε, ταυτόχρονα η πολυμορφία έχει αυξηθεί και επομένως θα πρέπει να δούμε το στοιχείο αυτό από πολύ πιο κοντά. Επίσης, προσπαθήσαμε να ε, δούμε συνθετικά και συνδυαστικά το πώς οργανώνεται η εργασία στην Ευρώπη και έχουμε βρει διάφορα προφίλ και διάφορες ομάδες ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το θέμα μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά κάποιες ομάδες. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία να τα γνωρίζουν καλά όσοι λαμβάνουν αποφάσεις. Πριν σας παρουσιάσω ε, την, τους αδείκτες ε, για την ποιότητα της απασχόλησης, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημαντικές διαστάσεις ή στοιχεία Πρώτον είναι ο διαχωρισμός αναφύλο. Γνωρίζουμε ότι αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να ε, πάρει διάφορες μορφές. Έχει υπάρξει κάποια πρόοδος ε, γνωρίζουμε λοιπόν ότι πλέον υπάρχουν και αρκετοί νεαροί άνδρες οι οποίοι παρέχουν αμυστή ε, εργασία, αλλά η απλήρωτη εργασία παραμένει ε, με γυναικείο πρόσημο στο μεγαλύτερο ποσοστό της. Επίσης ε, σε υψηλές θέσεις βρίσκονται περισσότερο άντρες παρά γυναίκες. Μονάχα 33% των εργαζομένων έχουν ως επικεφαλής γυναίκες. Επίσης μόνο το 21% των ε, θέσεων ε, μπορούμε να πούμε ότι ε, παρέχουν μια αρκετά, έναν αρκετά μεγάλο βαθμό ανάμειξη ανδρών και γυναικών. Εδώ σας δείχνω την εικονογράφηση των εργαζομένων βλέπετε ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανά κράτος μέλος και αυτό έχει επίπτωση στις ε, διαπραγματεύσεις ε, ε, με εργασιακά θέματα και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι διαπραγματεύσεις αυτές. Σύμφωνα με την έρευνά μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εκπροσώπηση των εργαζομένων και αυτό συμβάλλει πολύ στην βελτίωση της ποιότητας εργασίας. Τώρα, Όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, πρέπει να σας πω ότι έχουμε έναν δίκτυο, ο οποίος αναφέρεται ακριβώς στην εργασία. Προσπαθούμε ε, μέσω όλων των διαθεσίμων πληροφοριών να εξάγουμε την ε, πληροφόρηση η οποία αφορά ε, την ίδια την εργασία. Εμείς εστιάζουμε στην εργασία γιατί αυτό είναι το επίπεδο ε, το συμβατικό μεταξύ της εταιρείας και του ε, ατόμου. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό επίπεδο. και σε αυτό έχουμε τη δικαιοδοσία να ε, παρέμβουμε. Δεύτερη πληροφορία είναι να χρησιμοποιούμε όλες τις πληροφορίες ε, σχετικά ε, με την ε, ποιότητα. Δηλαδή, τι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη, τι είναι σημαντικό, τι πρέπει να συνυπολογιστεί έτσι ώστε να εκτιμηθεί η ποιότητα της εργασίας. Ξέρουμε πλέον ε, ως ε, τεκμήριο των ερευνών που έχουν γίνει ε, και είναι πολλές ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στη βελτίωση επιδείνου της υγείας με μια καλή ποιότητα ή όχι θέση εργασίας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία βέβαια. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι κάθε δείκτης βασίζεται σε 13 ε, υποδείκτες ε, εκτός από το ε, στοιχείο των αμοιβών. Μπορεί δηλαδή να ληφθούν υπόψη διαφορετικά στοιχεία σε κάθε περίπτωση έτσι ώστε να φτάσουμε από τις πιο γενικές και αφηρημένες πληροφορίες σε πιο συγκεκριμένα. Σε γενικέ γραμμέ μπορούμε να πούμε ότι όσο καλύτερο, όσο ψηλότερο είναι ο δείκτη τη ε, ποιότητα, ε, τόσο καλύτερα είναι και οι υπόλοιποι δείκτε εκτό από την ε, εντατικοποίηση τη εργασία. Επίσης ε, να πω ότι κάποιοι δείκτες ε, ε, περιέχουν μόνο θετικά στοιχεία, άλλοι στοιχεία θετικά και αρνητικά και επομένως δεν πρέπει κανείς να βλέπει την, τις τιμές, θα πρέπει να δει κανείς τις, τους δείκτες αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές εντός των δικτών. Εδώ έχω λοιπόν σε αυτή τη διαφάνεια 7 δείκτες ενώ στην επόμενη διαφάνεια, στην επόμενη διαφάνεια λέω, δείχνουμε ε, τις ε, τάσεις ε, επί τεσσάρων διαστάσεων και τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι έχουν υπάρξει βελτιώσεις όσον αφορά τις δεξιότητες. Όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν ας πούμε ε, κομπιούτερ, ε, υπολογιστές και επίσης ε, όλο και, περισσότερο, όλο και περισσότερα αιτήματα για κατάρτιση σημειώνονται. Ε, η μείωση της ε, έντασης ε, της εργασίας οφείλεται στο ότι έχουμε πολύ περισσότερες εναλλακτικέ, ας πούμε μορφές εργασίας. Όσον αφορά τις αλλαγές, είναι πολλές, μπορεί να αφορούν την ίδια τη δομή της απασχόλησης, μπορεί να, ε, να σημαίνει βελτίωση της προσωπικής εργασίας, ε, αλλά βεβαίως όσον αφορά τη διάρθρωση της απασχόλησης, η κρίση έπαιξε σημαντικό ε, ρόλο. Η εντατικοποίηση της, ή η ένταση της εργασίας ε, βλέπουμε ότι, το 2000, ε, ε, ότι από το 2005 στο 2010 είχαμε μείωση, αλλά από το 10 και μετά ξανά έχουμε και αυτό ήταν καλό νέο. Έκτοτε όμως έχουμε ξανά αύξηση των ποσοστών και αυτό δεν είναι καλό. Επίσης διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ε, διαφορετική εξέλιξη και μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά ε, το σημείο αυτό. Θα ήθελα τώρα να αναλύσω τα στοιχεία του κάθε δίκτυ ένα-ένα. Εδώ σας δείχνω μια διαφάνεια σχετικά με τις απολαβές. Εμείς χρησιμοποιούμε το πραγματικό επίπεδο ε, των ε, αμοιβών για να αναπτύξουμε αυτούς τους δείκτες επιότητας απασχόλησης θα πρέπει ε, να δούμε αξιολογήσεις όπου γίνονται μέσω αντικειμενικών στοιχείων. Τώρα, η πληροφορία η υποκειμενική ε, σχετικά με το κατά πόσον θεωρούν ότι είναι σωστή και δίκαιη η πληρωμή τους, ε, ε, θεωρούν οι ίδιοι εργαζόμενοι και αυτό συμπεριλαμβάνεται όμως. Φυσικό περιβάλλον είναι ο επόμενος δείκτης. Αυτός είναι ένας δείκτης για τον οποίο από το 1991 ήδη έχουμε στοιχεία. Ε, τα στοιχεία που έχουμε έδειξαν ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία ε, αύξηση ε, στους εργαζόμενους οι οποίοι χειρίζονται, οι οποίοι χειρίζονται χημικά, οι οποίοι χειρίζονται ανυψωτικά μηχανήματα ή που καλούνται να σηκώσουν βάρη οι ίδιοι. Επόμενος δείκτης όσον αφορά την ένταση της εργασίας για μας ε, που είμαστε ερευνητές ε, αυτό, ε, αυτός είναι ένας από τους δείκτες που μας απασχολούν περισσότερο. Ένταση εργασίας λοιπόν προκύπτει όταν δουλεύουμε με γρηγορότερους ρυθμούς, όταν γίνεται πιο πυκνή η εργασία. Επίσης όταν ε, ε, πρέπει ταυτοχρόνως να αντιμετωπίσουμε διαφορετικούς ρυθμούς και επομένως να πρέπει να διαλέξουμε τι είναι πιο επίγον και τι είναι λιγότερο επίγον, όταν δηλαδή ε, δεν, όταν έχουμε στενά περιθώρια. Ένα άλλο στοιχείο είναι είναι καταστάσεις οι οποίες ε, μπορεί συναισθηματικά να είναι πιεστικές ε, ή ενοχλητικές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον εργαζόμενο. Επίσης, όσον αφορά ε, τις ε, ποσοτικές απαιτήσεις, ε, οι τεχνίτες, οι χειρόνακτες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις. Απ' την άλλη πλευρά, όσο ανεβαίνουμε στο επίπεδο της απασχόλησης, οι δείκτες λίγο αλλάζουν. Ποιότητα χρόνου εργασίας. Εδώ θέλω να πω ότι ο μέσος όρος ορών εργασίας ε, ακολουθεί φθήνουσα πορεία, είναι μια τάση παλαιότερη η οποία, παλαιότερη, η οποία επιβεβαιώνεται ε, διαρκώς. Και επίσης ε, να σας πω ότι 22% των εργαζομένων ε, έχουν ε, ε, δηλώσει ότι δουλεύουν και στον ελεύθερο χρόνο τους έτσι ώστε να ολοκληρώσουν την εργασία που τους έχει ζητηθεί. 12% των εργαζομένων δηλώνουν ότι πολύ συχνά στη διάρκεια του μήνα αναγκάζονται να δουλέψουν με προειδοποίηση της τελευταίας στιγμής. Είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε ασάφεια των ορίων στην ε, Ευρώπη. Έχουμε ε, επίσης ε, πολλές εμπειρίες όσον αφορά την ευελιξία και την διαπραγμάτευση της ευελιξίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε πάνω στο θέμα αυτό. Ένα πέμπτος παράγοντας είναι το κοινωνικό περιβάλλον. Εδώ λοιπόν έχουμε θετικά στοιχεία, την κοινωνική υποστήριξη από τους συναδέλφους, από τους διευθυντές, Έχουμε επίσης και τα θέματα ηγεσία, διαχείρισης και διευθυντικών ικανοτήτων, σε τι βαθμό μας βοηθούν να κάνουμε τη δουλειά μας, να αναπτυχθούμε. Έχουμε δε και αρνητικούς δείκτες, αρνητικούς παραγοντές. Και βλέπετε εδώ στη διαφάνεια, σας παρουσιάζουμε αυτό που ονομάζουμε αρνητική κοινωνική συμπεριφορά. Περιστάσεις, για παράδειγμα, και περιπτώσεις βίας στον εργασιακό χώρο Τέτοια προστατικά αναφέρονται από 15% των εργαζομένων. Εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους. Και αυτό αποτυπώνεται κυρίως σε θέματα υγείας, δημόσιας διοίκησης και μεταφορών. Αυτό έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και υπάρχουν και σημαντικοί, σημαντικές πρωτοβουλίες για κοινωνικό διάλογο προς την κατεύθυνση. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε μια μεγάλη επιτυχία. Τα δεδομένα μας καταδεικνύουν ότι υπήρχαν κάποιες ε, επιτυχίες και βελτιώσεις με την πάρτα του χρόνου. Θα πρέπει παρόλα αυτά να σημειώσω την εξή απόχρωση. Καταρχάς, έχουμε 10% των εργαζομένων ακόμα, 21 εκατομμύρια δηλαδή εργαζόμενους, που ζήτησαν ε, κατάρτιση αλλά δεν την έλαβαν. Η κατάρτιση αυτή χορηγείται κυρίως στους πιο εξειδικευμένους εργαζόμενους και στις πιο τυπικές μορφές απασχόλησης. Η διάρκεια της κατάρτισης είναι αρκετά σύντομη, γενικώ πως. Δίνεται έμφαση από το 1991 στην ευρωπαϊκή πολιτική προς την κατεύθυνση αυτή και έχει σημειωθεί πρόοδος. Βλέπουμε λοιπόν τώρα τα prospects, οι προοπτικές. Τρία στοιχεία επιτρέπετε μου να τονίσω. Καταρχάς, όταν ρωτάμε τον κόσμο αν είναι αυτοαπασχολούμενος ή μισθωτός, 1% απαντάει ότι δεν ξέρει. Άρα χρειάστηκε να αναπτύξουμε και να τροποποιήσουμε ένα ερωτηματολόγιο για να λάβουμε απαντήσεις από αυτού. Είναι σημαντικό, θεωρώ αυτό. Σημαντικό πόρισμα αυτό. Κατά δεύτερον, αν κοιτάξουμε τους αυτοπασχολούμενους χωρίς τους μισθωτούς, ε, στην ομάδα αυτή διαπιστώνουμε ότι έχουν υπάρξει εξελίξεις και αλλαγές. Έχουμε αφενός τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι αυτοαπασχολούμενοι, αλλά με χαρακτηριστικά στην εργασία τους που τους ε, προσωμιάζουν με τους μισθωτούς οικονομικά εξαρτώμενοι εργαζόμενοι, το οποίο αποτελεί ένα καθεστώς σε κάποιες ε, χώρες, αλλά σε άλλες όχι. Ύστερα, έχουμε από την άλλη άκρη τους αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται πραγματικά για τον εαυτό τους, έχουν ε, πολύ χαμηλό μισθό, μάλλον χαμηλά έσοδα και χαμηλά, χαμηλό ρυθμό ώρων απασχόλησης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τι μας λένε λοιπόν τα στοιχεία αυτά. Τι μας λένε αυτοί οι δείκτες. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία τέλεια δουλειά, προφανώς. Χρειαστήκαμε όλα αυτά τα δεδομένα για να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Πάντα υπάρχει λοιπόν ε, η καλή και η κακή πλευρά. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε κάθε δουλειά. και πάντα είναι πιο εύκολο να βελτιώσει κάποιες συνθήκε σε μια ομάδα και όχι μόνο του. Αν βελτιωθεί λοιπόν η ποιότητα της απασχόλησης, και εδώ είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το πόρισμα της ανάλυσης, άρα καταδεικνύει, καταδεικνύουν οι έρευνε το εξή. Ότι αν βελτιωθεί η ποιότητα της απασχόλησης, αν βελτιωθεί μία από τις διαστάσεις της απασχόλησης, βελτιώνει αυτό αυτόματα όλη την εμπειρία της ε, εργασιακής ζωής. Οι δείκτες που χρησιμοποιούμε για την ε, εργασιακή ζωή είναι πολλαπλή. Άρα η ποιότητα της απασχόλησης έχει να κάνει με την καλύτερη υποκειμενική ευημερία, ευτυχία, με την ε, υγεία, λιγότερες απουσίες και ασθένειες με την αίσθηση ότι κάνει κανείς ε, χρήσιμη δουλειά, ωφέλιμη δουλειά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το να τα βγάζει πέρα κανείς σε οικονομικά ε, με τη δέσμευση, με τα κίνητρα, με το καλύτερο κοινωνικό και εργασιακό κλίμα, με καλύτερη ισορροπία εργασιακή και προσωπική ζωή. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πλεονεκτήματα τη ποιότητα τη απασχόληση έχουν πολλές επιπτώσεις σε πολλούς κλάδους. Άρα είναι σαφές ότι η ποιότητα της απασχόλησης αποτελεί ένα σημαντικό μέσο άσκησης πολιτικής για μας. Τέλος, σας τα είπα όλα αυτά, αλλά σας είπα και για τους δείκτες πόσο καλή είναι, αλλά τι κάνουμε στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ποιότητα της απασχόλησης. Αυτό κατοχυρώνεται και στην ε, συνθήκη. Πώς απαντούμε λοιπόν στο θέμα αυτό προσπαθούμε με στατιστικές τεχνικές και με ανάλυση να ομαδοποιήσουμε κάποιες ε, δουλειές σύμφωνα με το επίπεδο της ποιότητας απασχόλησης. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πέντε ομάδες θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη με διαφορετικά προφίλ. Η πρώτη ομάδα, high flying, στην Ευρώπη. Εδώ Έχουμε θετικό πρόσημο σε όλες τις διαστάσεις, εκτός από την ένταση εργασίας και την ποιότητα ωραρίου. 22% των θέσεων απασχόλησης είναι στην ε, κατηγορία αυτή. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει αυτό που ονομάζουμε smooth running. Θετική, θετικό πρόσημο παντού. Εκτός από τα έσοδα και τις ικανότητες. 25% των θέσεων απασχόλησης. Τρίτη ομάδα, active manual, ενεργή χειρονακτική. Πολύ χειρονακτικές θέσεις εργασίας, απαιτούν μεγάλη σωματική προσπάθεια και εδώ έχουμε 22% των δουλειών, των ε, θέσεων απασχόλησης. Ύστερα έχουμε δύο ομάδες πιο αρνητικές. Η πρώτη είναι η υποπίεση ομάδα, under pressure, θετική διάσταση σε ό,τι αφορά τι ικανότητες, σε ό,τι αφορά τις προοπτικές και σε ό,τι αφορά τα έσοδα, αλλά σε ό,τι αφορά το κοινωνικό περιβάλλον, την ικανότητα διευθυντική και άλλες κοινωνικές συμπεριφορές, έχουμε εδώ μεγάλη αρνητική διάσταση, μεγάλη ένταση και λιγότερο λιγότερη ποιότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας. Και η πέμπτη ομάδα απλά είναι η φτωχής ποιότητας θέσεις απασχόλησης, όπου υπάρχει αρνητικό πρόσημο σε όλους τους δείκτες. Πώς λοιπόν αυτά μπορούμε να τα συνδέσουμε και με την εργασιακή ζωή. Το μπλε, το χρώμα της Ευρωπαϊκής Σημαίας είναι το καλό, το θετικό και το πορτοκαλί είναι το αρνητικό. Τι διαπιστώνουμε λοιπόν στη διαφάνεια αυτή. Ότι ο κόσμος στις δύο πρώτες ομάδες, high flying και smooth running, αναφέρουν ότι είναι ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους σε ό,τι αφορά την ε, βιωσιμότητα της δουλειάς, την ισορροπία μεταξύ ζωής, προσωπικής και εργασιακής κτλ. Active manual, χειρονευτική ενεργή ομάδας αναφέρουν θετικές εμπειρίες, αλλά με ανησυχίες ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα. Οι άλλες δύο ομάδες αναφέρουν αρνητικές εμπειρίες από την εργασία και τη ζωή. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό ως πληροφορία, γιατί σύμφωνα με την πολιτική που θα αναπτύξουμε, Μάλλον, η πολιτική που θα αναπτύξουμε ενδεχομένως να έχει διαφορετικό αντίκτυπο στις διάφορες ομάδες εργασιών. Και αυτό φυσικά αφορά και τους στόχους της ανταγωνιστικότητας, της δέσμευσης και του καθεξής. Άρα, συνοψίζοντας, και έτσι δεν θα ξεπεράσει και το χρόνο που μου δώσατε, να θυμόμαστε το εξή. Η απασχόληση και το φύλλο παίζουν σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων. Υπάρχουν ανισότητες και διαστατικά ζητήματα τα οποία παίζουν μεγάλο ρόλο. Οι εθνικές πολιτικές και πρακτικές μπορούν να κάνουν τη διαφορά και μπορούμε να μάθουμε ημέρα από τους δε. Η ποιότητα της δουλειάς αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο συνδέεται με τη θετική εργασιακή εμπειρία. Μπορούμε να συζητήσουμε την κατεύθυνση που παίρνει η δουλειά του καθενός, αλλά με το που μπαίνουμε σε ένα θετικό κύκλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας στην Ευρώπη. Να βρούμε το συμβιβασμό. Να δούμε πώς μπορούμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση αμοιβαία επωφελή. Τα πλεονεκτήματα της ποιότητας της εργασίας αφορούν όχι μόνο τη ζωή του ατόμου, αλλά και πολλά, πολλούς άλλους παράγοντες, το είπα πολλές φορές αυτό, και διαφορά τα διαφορετικά πακέτα πολιτικής. Σύμφωνα με αυτά που θα συμφωνήσουμε να κάνουμε, αυτά που θα συμφωνήσουμε να κάνουμε, οι πολιτικές που θα αποφασίσουμε, θα έχουν διαφορετικό αντίκτυπο και θα πρέπει να σκεφτούμε εκ των προτέρων πώς θα επηρεαστεί η εργασιακή ζωή των ατόμων. Κάθε παράγοντας ε, της εργασίας μπορεί να βελτιωθεί μέσω πολιτικών και πρακτικών και η εκπροσώπηση των ε, εργαζομένων είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτεύξη καλύτερης ποιότητας της εργασίας. Και τέλος, πιστεύουμε πραγματικά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα της ποιότητας της ε, εργασίας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε πολύ για την ψηφιοποίηση, την παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι τέτοιου είδους μέσα Αξιολόγηση θα μας βοηθήσουν πολύ από πλευρά τη ανάλυσης και της έρευνας. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία, τα νούμερα, τα δεδομένα που μας δώσατε. Νομίζω ότι το είπαμε και στην εισαγωγή ότι η Eurofound είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη μέσων για να μετρηθεί η ποιότητα στην εργασία. Η πρώτη τέτοια έρευνα έγινε πριν από 25 ολόκληρα χρόνια. Έχει μεγαλώσει η έρευνα αυτή, έχει εξελιχθεί και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Γιατί αυτό το οποίο ακούμε είναι η άποψη των 44.000 ανθρώπων που απάντησαν για την έρευνα αυτή. Ο καθένας τους 45 λεπτά συνέντευξη έδωσε για να μας πει εμάς με λεπτομέρειες πώς έχει η δουλειά του, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας του και ζωής του. Και έτσι ερχόμαστε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη Θα καλέσουμε τώρα τους ε, Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους για να μας δώσουν εκείνη την άποψή τους όσον αφορά την βελτίωση της ποιότητας ηθικών εργασίας και γιατί έχει σημασία η βελτίωση αυτή. Λοιπόν, σας παρακαλώ, ο κύριος Βισεντίνη, η, η κυρία Ρενάτε Χορνουμτράους, ο κύριος Ντέβιτ Φόντεν, ο κύριος Κλοντρολά και ο κύριος Γιώργη Πυρίσκη. Παρακαλώ, ελάτε εδώ στο βήμα. Και ο Μισελ Σερβός, α, δεν είναι εδώ. Ίσως να μην τα καταφέρει να έρθει. Υπάρχει κάποιος που αντικαθιστά τον κύριο Σερβός εδώ. Ωραία, θα αρχίσουμε και θα δούμε αν θα έρθει τελικά. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όλοι εδώ. Χαίρομαι που σας έχω εδώ μαζί μου. Θα αρχίσουμε μπαίνοντα την ουσία του ζητήματος αμέσως. Όταν αρχίσαμε, ήτανε σαφές ότι αυτό που μετράει είναι το έργο της Eurofund και το έργο το δικό μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει αυτού. Και για προφανείς λόγους καταλαβαίνετε ότι σε καθημερινή βάση αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν με τους κοινωνικούς εταίρους, με την εμπειρία τους, τη γνώση τους, και είναι μια συνεχή συζήτηση, μόνιμη. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν και εμείς εδώ σήμερα θα συνεχίσουμε με το πρώτο τμήμα της συζήτησής μας για την ποιότητα της εργασίας. Έχουμε ονομάσει αυτό το τμήμα τη συνάντηση ποιότητα της εργασίας, προκλήσεις και ευκαιρίες. Ήθελε ο κύριος Σερβός να μας δώσει μια καλή εισαγωγή, αλλά αφού δεν είναι εδώ θα περάσουμε στους επόμενους. Να αρχίσω με τον κύριο Βισεντίνη, τι λέτε, που είναι ο Γενικός Γραμματέας της ETUC. Παρακαλώ, έχετε το λόγο και ενημερώστε μας για την ποιότητα εργασίας, προκλήσεις και ευκαιρίες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ήταν όντω πολύ ενδιαφέρον να ακούσω την παρουσίαση της έκθεσης πριν που πηγαίνει προς την κατεύθυνση και της δικιάς μας ανάλυσης. Αν και δικιά μας μερικές φορές είναι κάπως πιο απεσιόδοξη. Μάλλον γιατί εμεί έχουμε περισσότερο επαφή με τον χώρο, με τα μέλη μας. Τι βλέπουμε λοιπόν γενικά μιλώντας όσον αφορά την ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη. Βλέπουμε επιδείνωση της ποιότητας θέσεων απασχόλησης. Για δύο κύρια λόγους. Ο πρώτος είναι η οικονομική κρίση, γιατί δεν έχουμε βγει ακόμα από αυτή. Και η κρίση αυτή μας έφερε πολλές αρνητικές συνέπειες και επιπτώσεις στην ποιότητα της εργασίας, στις συνθήκες εργασίες και στην ζωή των ανθρώπων γενικά. Από την άλλη, οι διορθωτικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην αγορά εργασίας, αλλά και στους χώρους εργασίας, επίσης έχουν μερικές αρνητικές επιπτώσεις. Αν λοιπόν θα ήθελε κανείς να είναι ακριβέστερος, θα έπρεπε να εξετάσει τους 7 δείκτες, τους οποίους αναφέρατε και εσείς στην παρουσίασή σας, για να δούμε τι έχει γίνει στην πραγματικότητα για να δούμε κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε κάποιες από τις αρνητικές επιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα, προοπτικές. Αυτό έχει να κάνει με το καθεστώς εργασίας, δηλαδή με τη σύμβαση εργασίας που έχει κανείς. Έχει να κάνει με τη σταδιοδρομία, τις προοπτικές σταδιοδρομίας δηλαδή. Αλλά στη σημερινή κατάσταση πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με την προοπτική έβρεση εργασίας και διατήρησης της εργασίας. Δυστυχώς, επ' αυτού η κατάσταση είναι πάρα πολύ αρνητική και εμπιστοσύνη των ανθρώπων ότι θα βρούνε μια δουλειά ποιότητας και θα την κρατήσουν, η ελπίδα αυτή δυστυχώς είναι πάρα πολύ μικρή. Πάνω από 20 εκατομμύρια άνεργοι υπάρχουν στην Ευρώπη. Και ακόμα και αν τα τελευταία χρόνια ο κόσμος είχε κάποια ευκαιρία να βρει δουλειά γιατί κάποιες δράσεις εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη υπέρ της απασχόλησης, οι περισσότερες από αυτές τις ευκαιρίες είναι πολύ επισφαλείς. Μερικές φορές ατυπικές με μηδέν ώρες ε, σύμβαση, με κάτι άλλο. Δηλαδή, πολλά πρέπει να γίνουν προκειμένου να βελτιωθεί η αντίληψη και οι προοπτικές που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Ένα δεύτερο στοιχείο που μας απασχολεί είναι οι αμοιβέ. Από τα στοιχεία τα οποία έχουμε την τελευταία περίοδο, από διάφορα ο διάφορους διεθνείς οργανισμούς, όσα, διεθνές Τομείο κλπ. Σε όλες βασικά τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν μειωθεί οι μισθοί κατά μέσο όρο. Και οι μισθοί δεν ε, έχουν και προοπτικές. Και αυτό σε, όλες, σε όλες τις χώρες μέλη, ακόμα και στις χώρες μέλη εκείνες όπου η παραγωγικότητα έχει αυξηθεί, όπως είναι η Γερμανία ή η Πολωνία ακόμα, αλλά και σε χώρες όπως είναι η δικιά μου Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, όπου οι εξελίξεις στην παραγωγικότητα ήταν μηδαμινές. Παρ' όλα αυτά, ανάμεσα στην, ε, στις εξελίξεις στην παραγωγικότητα και τους μισθούς υπάρχει ένα χάσμα. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν για τα κέρδη των εργαζομένων και τις προοπτικές τους να έχουν μια καλύτερη δουλειά, καλύτερα πληρωμένη στο μέλλον. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσόντα ή δουλεύουν πιο εντατικά στη δουλειά που έχουν, συχνά πληρώνονται το ίδιο, όπως και παλιότερα. Σε μερικές περιπτώσεις έχουν και χαμηλότερες αμοιβέ. Αλλά αν πάμε στην κατηγορία των εργαζομένων που βρίσκονται στο πιο χαμηλό κομμάτι όσον αφορά τις δεξιότητες, τα προσόντα, την εντατική εργασία κλπ. Εκεί βλέπουμε πραγματική κατάρρευση των πραγματικών αμοιβών. Για το χρόνο εργασίας. Είδατε από τα στοιχεία ότι αυξάνει ο χρόνος εργασίας γενικά μιλώντας, αλλά πρέπει να αναλύσουμε γιατί. Επειδή υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία εργασίας προσωπικής ζωής, είναι επειδή με τον ίδιο μισθό οι άνθρωποι δουλεύουν ε, λιγότερο, υπάρχει περισσότερος αυτοματισμός, ε, ψηφιοποίηση. Ο χρόνος της εργασίας λοιπόν μειώνεται γενικά επειδή υπάρχει περισσότερη ανεργία, επειδή υπάρχει πιο επισφαλής εργασία και επειδή μικρά μονοκομμάτια της ε, εργασίας διαπιστώνουν αύξηση στον χρόνο εργασίας χωρίς βέβαια να συνάδουν και οι μισθοί. Πάντως γενικά έχουμε ε, μείωση του χρόνου εργασίας και μείωση και αμοιβών. Έρχομαι τώρα στις δεξιότητες. Πράγματι, σε κάποια τμήματα της αγοράς εργασίας υπάρχει ας πούμε επένδυση στην κατάρτιση των ανθρώπων στους χώρους εργασίας τους για να αυξηθούν τα προσόντα τους και δεξιότητέ τους. Αυτό όμως συμβαίνει μόνο για τις περιπτώσεις εργαζομένων υψηλού επίπεδου, δηλαδή υψηλών δεξιοτήτων και προσόντων. Στην χαμηλότερη γκάμα δεν ισχύει το ίδιο. Δεν υπάρχει κατάρτιση, ας πούμε, για όσους έχουν απολυθεί και προσπαθούν να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας ή για τους νέους που προσπαθούν για πρώτη φορά να βρουν μια δουλειά. Αν δείτε τις επενδύσεις που γίνονται ιδιωτικέ και δημόσιες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς τέτοιου είδους ε, επενδύσεις δεν υπάρχουν πια σχεδόν στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν επίγει να βρεθούν νέοι τρόποι για να γίνουν επενδύσεις στα προσόντα του εργατικού μας δυναμικού. Και δεν είναι σύμπτωση που βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε εκατομμύρια και εκατομμύρια ανέργους, έχουμε 1,2 κενέ θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Και δεν είναι δυνατόν να ταιριάξουμε αυτούς που δεν έχουν δουλειά με τις θέσεις απασχόλησης που είναι κενέ και υπάρχουν σήμερα στην αγορά εργασίας. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει μια αναντιστοιχία και οφείλεται στο ότι δεν γίνονται επαρκείς επενδύσεις στην κατάρτιση και την εκπαίδευση. Έχει υπάρξει επιδείνωση επίσης όσον αφορά την ασφάλεια, το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται κανείς. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες γιατί είναι πολύ περίπλοκη εικόνα. Η κατάσταση είναι περίπλοκη και όσον αφορά τα ρυθμιστικά πλαίσια που υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γίνονται βέβαια πρωτοβουλίες, αλλά η κατάσταση δεν έχει ακόμα βελτιωθεί. Και όσον αφορά το κοινωνικό περιβάλλον, όσο προχωράμε σε απορρίθμιση διαφόρων πλαισίων ασφαλείας, τόσο επιδεινώνεται και το κοινωνικό περιβάλλον. Οπότε, για τους κοινωνικούς εταίρους το θέμα δεν είναι μόνο να αναγνωριστεί πραγματικότητα, αλλά να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κενά, να τα καλύψουμε και να αντιμετωπίσουμε την τόσο αρνητική κατάσταση που διαπιστώνουμε στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Και πριν απευθυνθούμε στους θεσμούς να, για να ζητήσουμε να κάνουν κάτι, πρέπει πρώτα να κάνουμε εμείς κάτι. Και ο καλύτερος τρόπος είναι ο κοινωνικός διάλογος, οι κλαδικές σχέσεις, επιτόπου, στι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να κάνουν πολλά για να βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά βλέπετε, πρέπει να έχουμε στήριξη και βοήθεια από τις δημόσιες αρχές για να βελτιωθεί και η δικιά μας ικανότητα να βοηθήσουμε στις συλλογικές ε, ε, διαπραγματεύσεις, κάτι το οποίο δεν γίνεται σε πολλές χώρες σήμερα. Αντίθετα, επιδεινώνεται η ικανότητα κοινωνικών εταίρων να βοηθήσουν στις ε, κλαδικές αυτές σχέσεις. Από την άλλη, είναι σημαντικό να έχουμε και σωστές δημόσιες πολιτικές οι οποίες να αντιμετωπίζουν ένα-ένα τα 7 προβλήματα τα οποία εντοπίζει η έκθεση. Εμείς που είμαστε συνδικάτα βλέπουμε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά μας και είναι ο πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι κρίμα που ο Μισελ Σερβός δεν είναι εδώ σήμερα γιατί θα είχε περιγράψει πολύ καλά τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εφαρμοστεί ο πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Πάντως ο πυλώνα αυτός σίγουρα μπορεί να προσφέρει συγκεκριμένε ε, λύσει και γι' αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και θα πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Ενδεχομένω. Καλά θα κάνετε να περιοριστείτε σε 5-6 λεπτά. Και εσείς καλά θα είχατε κάνει να έχετε περιοριστεί σε 5-6 λεπτά, γιατί ιδάλλως θα έχουμε προβλήματα χρονικά. Αλλά αυτό ήταν δική μου ευθύνη. Έπρεπε να σας το είχα πει από την αρχή. Και τώρα να δώσω το λόγο στη Ρενάτε Ντράουσε. Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ε, Απασχόλησης στο Business Europe. Ευχαριστώ πολύ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ελπίζω να μου δώσετε και αντίστοιχες συνθήκες με τον συνάδελφο. Αντίστοιχο χρόνο, δηλαδή. Θα ήθελα καταρχάς να πω το εξής. Αυτή η μελέτη για τις ευρωπαϊκές ε, εργασιακές συνθήκες αποτελεί ένα από τα παραδοσιακά μέσα και μέσα για την κατάρτιση και τη χάραξη πολιτικής και για την ανάλυση που κάνει εδώ και κάποιο καιρό ε, το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Και καλημέρα και στον Μισελ, ο οποίος μόλις κατέφτασε. Και αυτό που θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το θέμα τώρα είναι η αντίληψη των εργαζομένων σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας. Και έχει σημασία αυτό. Προφανώ η αντίληψη μπορεί να διαφέρει σημαντικά και εξαρτάται και πάρα πολύ από την κουλτούρα. Και να χρησιμοποιήσω και το παράδειγμα του Λουκά, όταν κοιτάμε τον πίνακα με τους δείκτες ποιότητα ζωή του ΟΑΣΑ, ποιο είναι ο καλύτερο δείκτη σε ό,τι αφορά την αντίληψη μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ. Η απάντησή μου προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Γιατί προέκυψε ότι ο τρόπος που αξιολογούνται τα συστήματα υγείας από πλευράς του κόσμου είναι ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι έχουν ένα κακό σύστημα υγείας, ενώ οι Αμερικανοί θεωρούν ότι έχουν τα καλύτερα συστήματα υγείας. Και είναι μεγάλη η έκπληξη που μας πρόξενε λοιπόν αυτό το γεγονό και δείχνει το πώς η αντίληψη έχει σημασία και θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Υπάρχει η προσέγγιση λοιπόν της Eurofound που γίνεται συστηματικά εδώ και κάποια χρόνια και βλέπουμε ότι υπάρχουν αλλαγές σε ό,τι αφορά την αντίληψη, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι απασχαλούμενοι και οι αυτοπασχολούμενοι αξιολογούν τις εργασίες τους συνθήκες. Και εδώ θα ήθελα να πω το εξή. Και να σας πω το εξή ότι αυτή η έκτη έρευνα την οποία και συζητούμε τώρα καταδεικνύει ότι υπάρχουν ε, βελτιώσεις σε ό,τι αφορά τον τρόπο που γίνονται αντιληπτές οι εργασιακές συνθήκες. Και χαίρομαι και αυτό αποτελεί κάπως αντιστάθμισμα σε αυτά που λες εσύ Λούκα, που είπες ότι επιδεινώνεται η κατάσταση, αλλά εδώ τι βλέπουμε, ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι και έχει την αίσθηση ότι βελτιώνονται οι συνθήκε εργασία σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την έκθεση σε φυσικού κινδύνου, σε σημαντικού κινδύνου, σε ό,τι αφορά την ποιότητα των εργασιακών όρων. Και το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα για μένα είναι το εξή. Μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων, 85% συγκεκριμένα, είναι ικανοποιημένοι ή έως και πολύ ικανοποιημένοι με τις εργασιακές του συνθήκες. Είναι σημαντικό αυτό γιατί έχει αυξηθεί το ποσοστό από την έρευνα του 2000. Τότε ήταν 82% το ποσοστό αυτό. Άρα η αντίληψη που επικρατεί είναι ότι έχουν βελτιωθεί οι εργασιακές συνθήκες. Κάτι άλλο πολύ εντυπωσιακό. 81% των εργαζομένων αναφέρει ότι υπάρχει καλός συνδυασμός τη της κοινωνικής, οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική είναι κάτι το οποίο απαντά στα ζητήματα τα οποία υφίστανται. Και θα καλούσα λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το σκεφτεί αυτό πραγματικά. Να σκεφτεί την ανάγκη να υπάρξει ε, ένα συνεκτικό πακέτο για την ισορροπία μεταξύ εργασιακή και οικογενειακή ζωή, γιατί φαίνεται ότι μεγάλο ποσοστό, 80% δηλώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Να δούμε λοιπόν τι εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω και να υπογραμμίσω, το θέμα τη ποιότητα στην απασχόληση. Πρόκειται ένα θέμα το οποίο φυσικά οι εταιρείε από μόνε του και οι κοινωνικοί εταιρείε συνολικά το παίρνουν στα σοβαρά και υπάρχουν προφανώς μεγάλες προκλήσεις. Έχουμε το θέμα της κατάρτισης της εκπαίδευσης, την πρόκληση της οργάνωσης της εργασίας σε διαφορά την υγεία και την ασφάλεια. Έχουμε τη δημογραφική πρόκληση, αλλά ως κοινωνική εταίρη νομίζω ότι είμαστε περήφανοι που ε, τουλάχιστον τις ε, εξετάζουμε αυτές τις προκλήσεις, προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε, κοιτάμε την εργογύρανση, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους σε όλες τις χώρες, μαζί με το Συμβούλιο Εργασίας, τους εκπροσώπους των εργαζομένων, πώς μπορούμε να βρούμε, να βρούμε πολιτικές προκειμένου οι εργαζόμενοι να μείνουν στις θέσεις απασχόλησης πιο πολύ εφόσον το επιθυμούν και να υπάρχει πιο ομαλή μετάβαση. Έχουμε ένα πρόγραμμα εργασία επίση για την πτύχη της ψηφιοποίησης ό,τι αφορά την, ε, τον επαγγελματικό βίο. Και εδώ θα πρέπει να το συζητήσουμε. Ξέρετε, όλοι μιλάνε για την ε, ψηφιοποίηση, αλλά εμεί θα πρέπει να αναλύσουμε συγκεκριμένου παράγοντε. Τι είναι σχετικό και σημαντικό για μας από ευρωπαϊκή άποψη. Προετοιμάζουμε λοιπόν ένα σεμινάριο το οποίο θα λάβει χώρα του χρόνου το Φεβρουάριο, όπου και ελπίζουμε να έχουμε καλή αναρρετική χορήγηση στοιχείων από τους εμπλεκόμενους φορείς. Άρα, εγώ τι διαπιστώνω συνολικά, ότι η μελέτη καταδεικνύει ότι υπάρχουν και θετικές ε, εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας. Αυτή είναι η αντίληψη τουλάχιστον. Κάτι άλλο που είπες επίσης, Λούκα, για τους μισθούς και την αύξηση τους, τους πραγματικούς μισθούς που έχουν βελτιωθεί πιο πολύ από τις εργασιακές συνθήκες. Φυσικά, από μακροοικονομικής πλευράς, αν θέλει κανείς να δημιουργήσει ε, καλής, ε, μάλλον είπε ότι αυξάνονται λιγότερο οι μισθοί από την παραγωγικότητα. Φυσικά από μακροοικονομική πλευρά, αν θέλουμε να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τι θέσει απασχόληση, θα πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να αυξηθούν λιγότερο οι μισθοί σε σχέση με την παραγωγικότητα. Και στη Γερμανία γίνεται κάτι τέτοιο. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την απασχόληση και να ενταχθούν πιο πολλοί άνθρωποι στην αγορά εργασία, ο μοναδικό τρόπο να γίνει αυτό από μακροοικονομική πλευρά είναι να υπάρχουν ε, αυξήσεις μισθού που να επιτρέπουν πιο πολλές θέσεις απασχόλησης. Ε, το ξέρουμε στο οικονομολόγιο, δεν γίνεται όλα ταυτόχρονα. Αυτό το μικροοικονομικό φαινόμενο κάθε αυτό δεν είναι αρνητικό. Θα πρέπει να το αναλύσουμε. Άρα, θα έλεγα στο σημείο αυτό ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την ανάλυση και τους ε, παράγοντες που κρύβονται πίσω από αυτήν για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε συνολικά την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πολύ. Βλέπετε ότι πραγματικά εκφράζουν αυτό που εκφράζουν πάντα οι κοινωνικοί εταίροι. Και αυτό είναι εξαιρετικά καλό ε, ε, σημάδι και δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο κοινωνικός διάλογος και επίσης ότι είναι ακόμα ζωντανό πράγμα ο κοινωνικός διάλογος. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κυρία Σερβός από την Κομισιόν, από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Είστε Γενικός Διευθυντής σε αυτή την ε, Γενική Διεύθυνση. Ε, θα έπρεπε να είχατε ξεκινήσει εσείς σύμφωνα με το πρόγραμμα, αλλά παρόλα αυτά είμαι βεβαία ότι ε, και τώρα θα είσαστε σε θέση να μας πείτε την άποψή σας. Έχουμε ακούσει κάποια στοιχεία τα οποία μας δίνουν ελπίδα. Θα ήθελαμε τώρα να μοιραστείτε λίγη από τη γνώση σας μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη ε, που αργοπόρησα και λυπάμαι που δεν άκουσα ε, τα όσα είπε ο Λούκας πριν και η Ρενάτε μετά. Ε, καταλαβαίνω βεβαίως ότι ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη, βλέπει από τη δικιά του οπτική γωνία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι μου άρεσε ιδιαίτερος αυτή η έρευνα, ιδίω φέτος γιατί ε, δουλεύουμε υπό τον πυλώνα των κοινωνικών ε, δικαιωμάτων ε, και μας δίνει, λέω, τη δυνατότητα να απεικονίσουμε την πραγματικότητα της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα διδάγματα τα οποία μπορώ ε, να ε, συμπεράνω είναι τα εξής. Πρώτον, έχουν βελτιώσει έχουμε κάποιες βελτιώσεις. Ας πούμε, με ενδιαφέρον ε, διαπιστώνω ότι μεταξύ του 2005 και του 2015 έχει βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας και αυτό είναι πολύ θετικό. Βεβαίως αυτοχρόνως οφείλω να σημειώσω ότι ε, αυξάνεται και η περιπλοκότητα ε, τον, της απασχόλησης που αναφέρεται ε, περίπου σε αύξηση 50% τεράστια δηλαδή αύξηση αυτού και μόνο του στοιχείου. Αυτό απεικονίζει ε, την ε, εξέλιξη της εργασίας ε, στην έρευνα για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε χτες αναφέρεται κάτι αντίστοιχο ότι δηλαδή έχει γίνει πολύ περίπλοκη η πραγματικότητα αλλά εδώ κατανοούμε ότι αυτή η περιπλοκότητα αφορά πλέον όλα τα επίπεδα της, της απασχόλησης ε, και επίσης ότι οι μικρών δεξιοτήτων δεξιοτήτων, μικρών απαιτήσεων σε δεξιότητες θέσεις έχουν μετακυλήσει προς μεσαίες ε, ή ακόμα και ανώτερες, δηλαδή με μεγάλες απαιτήσει δεξιοτήτων. Δεύτερο στοιχείο είναι η, η σημασία της ισορροπίας της εργασιακής ε, ζωής. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό που σε τούτη την έρευνα ε, πλέον αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία σε τέτοιου είδους στοιχεία από ό,τι πριν. Οι σχέσεις είναι πλέον πιο περίπλοκες, οι, άνθρωποι προσπαθούν να συνδυάσουν όλο και περισσότερα πράγματα και αυτές οι καταστάσεις απαιτούν την ευελιξία συμφωνίας μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής και εμείς στην Κομισιόν θα πρέπει να το δούμε αυτό ε, και ενδεχομένω να αντιδράσουμε με κάποιες προτάσεις. Είναι προφανές ότι αυτή η μελέτη ε, ε, δείχνει και τα στοιχεία τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα. Ε, ας πούμε το, την ε, αυτοαπασχόληση. Από το 2013 έχουν δημιουργηθεί 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, ε, αλλά κυρίως αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους τέτοιου είδους θέσεις και επίσης ε, ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες, freelance, εργαζόμενοι σε συνθήκες υπεργολαβίας κτλ. Και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να δούμε γιατί είναι σημαντικά για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση αλλά είναι σημαντικά και για μας, για την αποστολή που έχουμε θέσει στους εαυτούς μας και πρέπει να αναρωτηθούμε το νομοθετικό πλαίσιο είναι κατάλληλο για να αντιμετωπίζει αυτό είναι την αλλαγμένη πλέον κατάσταση. Επίσης, ένα σημαντικό σημείο το οποίο σημειώνω είναι το θέμα των μισθών και συνδέεται βεβαίως οπωσδήποτε με την ποιότητα της εργασίας. Ναι, ε, υπάρχει ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας, επομένως ε, θα πρέπει ο μισθός να ευθυγραμμίζεται με την ανταγωνιστικότητα, έτσι ώστε να ε, συνεχίσει η δυνατότητα δημιουργίας απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά αυξημένος μισθός σημαίνει και αυξημένη εσωτερική ε, κατανάλωση. Θα πρέπει επομένω να βρεθεί ε, η σωστή ισορροπία. Η γραμμή της ε, Κομισιόν, αυτή στην οποία επιμένει, είναι ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη η οποία θα ακολουθεί και τα την ε, παραγωγικότητα ε, και προς τις δύο κατευθύνσεις δηλαδή και προς τα πάνω και προς τα κάτω ε, θα πρέπει να χρησιμοποιεί θα πρέπει ο καθένας στο επίπεδο λήψεων αποφάσεων να αναλάβει τις ευθύνες του. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω αφορά την κοινωνική προστασία. Αυτές οι νέες αναδυόμενες καταστάσεις καταδεικνύουν ότι υπάρχουν κάποιες ασυμμετρίες στον τρόπο παροχής ε, της ε, κοινωνικής ε, προστασίας σε διάφορες μορφές εργαζομένων και στους αυτοαπασχολούμενους και στους μισθωτούς. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν θέλουμε να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο λειτουργίας αγοράς θα πρέπει ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να παράσχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά την κοινωνική προστασία των ατόμων. Αυτά θέλω να πω ε, ε, ε, εκπροσωπώντας κατά κάποιο τρόπο τον πυλώνα της κοινωνικής προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Φόντεν, ο οποίος είναι τμήματάρχης στην Eurofound για τις ηθικές εργασίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουσα τις ε, παρουσιάσεις και θα προσπαθήσω να αντιδράσω κιόλα. Πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι στο επίπεδο που γίνεται η ανάλυση μας υπάρχουν μάλλον περισσότερα καλά νέα παρά κακά. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να αγνοούμε. Αλλά όπως είπε και η Ανιές, καμία θέση απασχόλησης δεν είναι τέλεια και υπάρχουν και θύλακε όπου εκεί δυστυχώς βλέπουμε πολλές αδυναμίες σε πολλές διαστάσεις. Άρα σίγουρα έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά ακόμα. Τώρα, να απαντήσω λίγο στα σχόλια της Ρενάτε, κάπως σύντομα, για τις αντιλήψεις. Τι εννοεί κανείς αντιλήψεις. Στην ε, ανάλυση μας πάμε στους εργαζόμενους, γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί είναι οι πιο κατάλληλοι να μας μιλήσουν για τις συνθήκες εργασίας τους και για τη ζωή τους. Και κάνουμε ερωτήσεις που βέβαια επιδέχονται υποκειμενικές απαντήσεις και τις χρησιμοποιούμε, αλλά υπάρχουν και δείκτες για την εκπόνηση πολιτικής και αυτοί οι δείκτες έχουν να κάνουν μόνο με τις αντικειμενικές ερωτήσεις και απαντήσεις. Περισσότερο με την υγεία. Οπότε, ναι, υπάρχουν κάποια υποκειμενικά στοιχεία στην έκθεσή μας, αλλά δεν πρόκειται για αντιλήψεις. Προσπαθούμε όσο γίνεται καλύτερα να απεικονίσουμε την πραγματικότητα στη μελέτη μας. Το άλλο γενικό που θέλω να πω είναι ότι συζητάμε διάφορα επίπεδα. Έχουμε ακούσει για τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, πώς βοηθούν στις διαπραγματεύσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον κοινωνικό πυλώνα. Υπάρχουν κοινωνικές πολιτικές, η νομοθεσία, οι... τις διακρίσεις στις διάφορες χώρες μέλη. Αλλά αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι και το τοπικό επίπεδο, το επίπεδο της επιχείρησης, γιατί υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που κρατούν το κλειδί της πραγματικότητας και διαμορφώνουν την πραγματικότητα. Επιχειρήσεις όπου είναι με τους κοινωνικούς εταίρους που αποφασίζονται τα ωράρια εργασίας, η διαχείριση των χώρων κλπ. Και αυτά είναι αποφασιστική σημασίας σε ένα μεγάλο βαθμό για τις ηθίκες εργασίας. Συνεπώς, πώς διαρθρώνονται τα διαφορετικά επίπεδα και πώς συνδυάζονται οι δράσεις των κοινωνικών εταίρων με τη δράση των πολιτικών αρχών σε διάφορα επίπεδα. Θέλω όμως τα λίγα λεφτά που μου μένουν να αναφερθώ σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Το ένα είναι οι δεξιότητες και τα προσόντα. Μεγάλη ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Σε διεθνές επίπεδο αυτή η αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα και τις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης. Ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα στην ε, έρευνά μας είναι ότι το 40% των εργαζομένων λένε ότι θα έπρεπε να έχουν περισσότερη κατάρτιση για να κάνουν τη δουλειά τους και δύο φορές τόσοι λένε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντά τους. Εδώ σημαίνει ότι διαθέτουμε ένα τεράστιο δυναμικό και για να επανέλθω στο επίπεδο της επιχείρησης εξαρτάται από τον σχεδιασμό των θέσεων εργασίας και από το επίπεδο δράσης και κατάρτισης. Δεύτερον, ένα άλλο παράδειγμα που το ακούσαμε και στην παρουσίαση. Ναι, υπάρχει πρόοδος όσον αφορά τις διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων και πώς θα ανεβαίνουν πιο ψηλά οι γυναίκες. Παρόλα αυτά, οι γυναίκες διαχειρίζονται μικρότερες ομάδες, ή ομάδες γυναικών κυρίως. Οπότε ο διάβολος βρίσκεται στη λεπτομέρεια θα έπρεπε να σκαλίσουμε περισσότερο εδώ την έρευνα. Συνεπώς, ναι, υπάρχει πρόοδος και αρκετά καλά νέα, αλλά να μην ξεχνάμε και να μην αγνοούμε την όλη ιστορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Κλοντ Ρολάν, που είναι Ευρωβουλευτής, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πρώτα από τη δικιά μου πρακτική και την εμπειρία που έχω τη συνδικαλιστική. Γιατί 40 χρόνια αυτή ήταν η δουλειά που έκανα. Και βάσει αυτού παρεμβαίνω και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε 40 χρόνια λοιπόν μπορώ να σας πω ότι έχω δει τεράστιες αλλαγές και τεράστια εξέλιξη όσον αφορά τις ηθικές εργασίας. Αρκεί να κοιτάξει κανείς ποιο ήταν το περιεχόμενο των συλλογικών συμβάσεων πριν από 40 χρόνια που ανέφεραν τη φυσική ασφάλεια, το χρόνο εργασίας, τις αμοιβέ. Τίποτα άλλο. Σήμερα ακόμα υπάρχει αυτή η προβληματική βέβαια, παρούσα, αλλά έχουν προσθεθεί και πολλά άλλα στοιχεία. Έχουμε αυξήσει τα στρώματα Κυρίως μιλάμε για την ποιότητα της ζωής στην εργασία, αλλά και την ποιότητα της ζωής γενικότερα. Γιατί οι μισθωτοί δεν ε, είναι άνθρωποι μόνο όταν δουλεύουν, έχουν και μια δουλειά εκτός εργασίας. Μια, συγγνώμη, ζωή εκτός εργασίας. Οπότε τι μαθαίνουμε όσον αφορά αυτή την ποιότητα ζωή, ότι επιδεινώνεται. Ότι οι εργαζόμενοι θα την ήθελαν καλύτερη, θα ήθελαν καλύτερες συνθήκε μεθαύριο. Πώς θα συνδυάσουμε το χρόνο που θα αφιερώσουμε στην οικογένεια, στον ιδιωτικό βίο, στην εργασία. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα και εδώ θα αντιδράσω λίγο στην ε, συνάδελφο που λέει ότι οι περισσότεροι λένε δεν υπάρχει πρόβλημα συμφιλίωσης. Ε, λοιπόν, στις επιχειρήσεις που εγώ ασχολήθηκα με τα παιδιά, για παράδειγμα, δεν υπήρχε πρόβλημα. Γιατί? Γιατί αφού έτσι καλώς δεν υπήρχε τίποτα, δεν είχε προβλεφθεί τίποτα, ε, οι μισθωτοί αυτόνομα έπρεπε να βρουν λύσεις με τους παππούδες, τους φίλους, τους γείτονες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Επίσης υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας στην απασχόληση. Ο φόβος δηλαδή ότι κανείς θα χάσει ίσως τη δουλειά του αλλάζει την αντίδρασή τους. Η επισφαλής εργασία επίσης αλλάζει τη συμπεριφορά και όλα αυτά οδηγούν στον κοινωνικό διάλογο να υπάρξει διαφορετική δράση από πλευρά των υπευθύνων. Ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει, ο φόβος ε, υπερισχύει και έτσι τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά. Τώρα, κάτι που ήθελα να προσθέσω είναι μια σύγκριση στην Ευρώπη όσον αφορά την απουσία από την εργασία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό για να εντοπίσουμε τη διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την ποιότητα στην εργασία. Φυσικά, ανάλογα με τους κλάδους, επιχειρήσεις κτλ. υπάρχουν διαφορές, ανάλογα με τις περιοχές και την ανεργία, αλλά από την μελέτη αυτή που είδα, εγώ είδα ότι υπάρχουν τρεις καθοριστικοί παράγοντες από ό,τι φαίνεται όσον αφορά την απουσία από την εργασία και τη δυνατότητα κινητοποίησης των εργαζομένων. Είναι η αναγνώριση, το νόημα της δουλειάς που κάνει και η συλλογικότητα. Αυτά τα τρία στοιχεία είναι πολύ σημαντικά. Και για παράδειγμα, όσον αφορά το νόημα τη εργασία, όταν βλέπουμε διάφορε έρευνε για του νέου, τι λένε οι νέοι εργαζόμενοι. Λένε θέλω δουλειά, αλλά θέλω μια δουλειά η οποία να δίνει κάποιο νόημα στη ζωή μου. Να έχει νόημα. Και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Και το τελευταίο από την έρευνα αυτή είναι η μακρά σταδιοδρομία. Όσο προχωράμε στην ηλικία, τόσο πιο συχνά λείπουμε από τη δουλειά. Και όσο υπάρχουν πολιτικές που αυξάνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, θα έχουμε όλο και περισσότερο πρόβλημα με την απουσία από την εργασία. Για μένα λοιπόν η πρόκληση, είναι πρόκληση και για τις επιχειρήσεις και για τους μισθωτούς και για τους πολιτικούς. Η πρόκληση είναι λοιπόν κάπου να συντονιστούν όλα αυτά στην εργασία, λαμβάνοντας υπόψη νέα στοιχεία. Το θέμα του φύλου για παράδειγμα. Οι παράγοντες ε, στρες που οδηγούν σε βία στην εργασία και στην ε, παρενόχληση. Όλα αυτά είναι καθοριστικά. Επίση, όταν γίνονται αλλαγέ, γιατί στις επιχειρήσεις γίνονται αλλαγέ πολύ πιο γρήγορα σήμερα από, το παρελθόν. Θα έπρεπε να είναι προβλέψιμες αυτές οι αλλαγέ, να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για να προσαρμοστούν καλύτερα. Και υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας. Μιλήσαμε για ευελιξία. Σίγουρα είμαστε σε ένα κόσμο πολύ πιο ευέλικτο. Όμως πρέπει η σταδιοδρομία του καθενός να εξασφαλίζεται. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Η ποιότητα της ζωής μειώνεται. Έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διάφορες ιδέες. Μπορεί να ακούγεται σλόγγαν, αλλά όταν λέει ο Γιούγκερ ότι θέλει το τριπλό α και στην κοινωνική Ευρώπη, γίνεται με τον κοινωνικό διάλογο, τον κοινωνικό πυλώνα, όλα όσα βρίσκονται στο τραπέζι σήμερα και συζητάμε εδώ στην Επιτροπή μας, είναι αυτά η οδηγία για τους απασπασμένους, την αδήλωτη εργασία. Εσύ κάνεις έκθεση, έτσι, η συγκήτρια για τα καρκινογόνα, τις καρκινογόνες ουσίες. Εδώ και καιρό δεν το είχαμε ασχοληθεί αυτό το ζήτημα, είναι καλό που το κάνουμε τώρα. Συνοψίζοντας λοιπόν, για μένα, το πρώτο είναι η απασχόληση, το μέγεθος της απασχόλησης, ποσοτική έκφραση. Το δεύτερο είναι να προλαμβάνουμε τις αλλαγές, να τις προβλέπουμε και να συμμετέχουμε σε αυτές. Και το τρίτο είναι ο κοινωνικός διάλογος στην επιχείρηση, ο κοινωνικός διάλογος στους κλάδους και ο κοινωνικός διάλογος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε τα μέσα στη διάθεσή μας. Η Επιτροπή απασχόληση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα τέτοιο μέσο και εδώ δίπλα έχουμε και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Αυτό που με ενδιαφέρει πολύ, γιατί νομίζω πολλά ενδιαφέροντα γίνονται στον κόσμο εργασία. Είδα τα αποτελέσματα μια μεγάλη έρευνα για την εργασία που έκανε η CFDT στη Γαλλία. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα δυναμική, στην οποία καλό θα ήταν να σταθούμε για την αυριανή απασχόληση, πώς εξυγχρονίζεται, πώς ψηφιοποιείται, τι, πώς αλλάζει. Και στην Επιτροπή ξέρω ότι υπάρχει μια τέτοια προβληματική. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και θα τελειώσω, όχι θέλοντας να κολακέψω κανέναν, γιατί είμαστε εδώ με τον ε, Φόντεν, αλλά να ξέρετε ότι για μας αποτελείται κάτι το πολύτιμο. Είναι ζωτική σημασία να μπορούμε να στηριχτούμε στο δικό σας έργο, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εμεί τη δουλειά μας εδώ στο Κοινοβούλιο, αν δεν μπορούσαμε να βασιστούμε στη δικιά σας ε, δουλειά, στη δουλειά οργανισμών όπως είναι το Eurofound. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι είναι όπως τα είπατε ακριβώς. Δηλαδή εμείς αποδίδουμε μεγάλη σημασία ε, στις ερωτήσεις, όχι απαραίτητα στις ε, απαντήσεις. Και οπωσδήποτε σίγουρα στο, ε, στην Eurofound αποδίδουμε μεγάλη σημασία η οποία θέτει τις ερωτήσεις και οι οποίες μας δείχνουν ακριβώς τι γίνεται ε, στην ε, Ευρώπη. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Επενδύση ο οποίος επίσης είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσωπεί την ομάδα ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Όπως ε, ανέφερε και ο κύριος Ρούλαν προηγουμένως, έχετε ενεργά εμπλακεί ε, με το θέμα της αδήλωτης εργασίας. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, αλλά βεβαίως σας δίνω το λόγο. Είμαι ιδιαίτερο ευτυχή που συμμετέχω σε αυτό το πάνελ, οφείλω να ομολογήσω. Θα προσπαθήσω να συμβάλλω σε αυτό το γενικότερο ζήτημα που αποτελεί και το στόχο ε, τέτοιων συζητήσεων, δηλαδή ποιε είναι ή ποιε μπορεί να είναι οι συστάσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ο ήδη έκανε τρει συστάσει. Πρώτα απ' όλα όμω να πω ότι από την, ε, όσον αφορά την ε, έρευνα η γενική εντύπωση πέρα από το κατά πόσον υπάρχει ε, βελτίωση ή όχι, ε, είναι ότι κανείς μπορεί να δει το ποτήρι είτε μισοάδιο είτε μισογεμάτο. Ακούσαμε ε, διαφορετικές εκτιμήσεις όσον αφορά αυτό το περίπλοκο θέμα. Οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις οι οποίες είναι παρούσες, αλλά, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχουν και ζητήματα τα οποία μας προκαλούν μέγα προβληματισμό. Εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα έβριμα το οποίο πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο αντικατοπτρίζει κάποιο, ένα πολύ χαρακτηριστικό ε, στοιχείο που αφορά τάσεις, εν πάση περιπτώσει, αν όχι τελικό στοιχείο. Αναφέρομαι σε ένα έβριμα συγκεκριμένο. Δηλαδή ότι η αναλογία εργαζόμενων που θεωρεί ότι η εργασία που είναι καλά καμωμένη έχει μειωθεί από το 51% το 2005 στο 45% στο 2010 και 40% το 2015. 5% των εργαζομένων ποτέ ή σπανίως έχουν την αίσθηση ότι έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Ο κύριος Μενέντες Βάλτες ε, στην αρχική του παρέμβαση σήμερα το πρωί διασύνδεσε το θέμα της ε, ποιότητας ε, της απασχόλησης ε, με την παραγωγικότητα. Οι δε συμμετέχοντες στο πάνελ, ο καθένας από την δικιά του άποψη συνέδεσαν το θέμα και με τις ευκαιρίες απασχόλησης και με την αμοιβή. Κατά τη δική μου άποψη, εάν θέλουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα, και αν θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη, είναι να κάνουμε ό,τι γίνεται περισσότερο έτσι ώστε να απασχοληθούν ε, οι άνθρωποι με τον ε, πιο παραγωγικό τρόπο. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία είναι ατέρμον. Ε, δηλαδή από τη μία η κοινωνική πρόοδος, κοινωνική προστασία και από την άλλη η παραγωγικότητα. Αλλά εδώ έχουμε μια κατάσταση, πρέπει να έχουμε μια κατάσταση win-win. Εδώ έχουμε πληθώρα ε, στοιχείων στην έρευνα αυτή και φαίνεται ότι στοιχειων στην ερευνα αυτη και φαινεται οτι παραμενει ένα μεγάλο ποσοστό παραγωγικότητας το οποίο δεν καταφέρνουμε να ενεργοποιήσουμε, να κινητοποιήσουμε. Αυτό είναι το ένα μου σημείο. Και βεβαίως εδώ θέλω να συμφωνήσω με αυτούς που είπαν ε, ότι πίσω από την γενική ιδέα ε, της ε, μέσης ποιότητας ε, ε, απασχόλησης, ε, της ποιοτικής απασχόλησης κτλ που βεβαίως όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, ε, κυρίως σε μια εποχή που η ασταθής εργασία ε, αυξάνεται Ε, ε, εξεκολουθούμε να θεωρούμε την ποιότητα της εργασίας ένα σημαντικό θέμα ε, και αυτό το πολύ σοβαρό και ιδιαίτερα, ιδιαίτερα ανησυχητικό θέμα της μη ασφαλούς εργασίας πραγματικά αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το μέλλον γιατί αποτελεί μεγάλη απειλή. Ειδικά αν το δούμε από κοινού με την ψηφιοποίηση και άλλες εξελίξεις. Επίσης παραμένει το μεγάλο κεφάλαιο και η μεγάλη πρόκληση ε, των ανισορροπιών και των ανισοτήτων ε, στους πίνακες τους οποίους μας δείξατε ε, προκύπτουν αυτές οι ανισότητες. Μιλισμονούμε ότι οι ανισότητες αυτές ε, κοστίζουν, έχουν ένα κόστος σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ε, απασχολούνται ε, οι εργαζόμενοι, όσο αυξάνονται οι ανισότητες, αυξάνονται οι τριβές και οι συγκρούσεις. Ε, Βεβαίω καταλαβαίνω ότι, ότι μετά θα έχουμε τη δυνατότητα ε, να έχουμε ερωτήσει και απαντήσεις και ενδεχομένω τότε θα ακούσουμε ε, και από τους άμεσα ενδιαφερόμενους για κάποια θέματα τα οποία σχετίζονται με το θέμα αυτό. Αλλά το ζήτημα των ανισοτήτων, το ζήτημα της φαιάς οικονομίας που διαβρώνουν τις βασικές αρχές ε, της υγιού, του υγιούς ανταγωνισμού και των καλών θέσεων, των ποιοτικών θέσεων εργασίας, είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και μάλιστα πρέπει να πω ότι είναι προβλήματα αυτά που έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις σε μερικές χώρες. Τέλος, ο κύριος Σαρβός αναφέρθηκε στην ε, ετήσια ε, έκθεση για την ανάπτυξη η οποία ε, υιοθετήθηκε χτες. Και είναι σημαντικό ε, που η Κομισιόν πλέον ε, δείχνει ενδιαφέρον σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα των, των κοινωνικών προβλημάτων και του κοινωνικού πυλώνα. Και εγώ θεωρώ ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και ότι σοβαρή δουλειά πρέπει να γίνει. Ε, εδώ βλέπω ότι ε, γράφεται και μία σειρά ε, κεντρικών σημείων που απαιτούν ανταπόκριση και από την Ευρώπη. Βλέπουμε, ας πούμε, την φορολογική η πολιτική, βλέπουμε την κοινωνική πολιτική, βλέπουμε ένα σωρό στοιχεία, χρηστή διαχείριση. Ωραία, τα καταλαβαίνω αυτό, ε, ο κύριος ε, Σαρβός αναφέρθηκε στους ίδιους τους ε, κανόνες και αναρωτήθηκε κατά πόσον οι κανόνες που υπάρχουν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις νέες αλλαγμένες συνθήκες. Ε, τώρα το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δούμε ε, και τις ίδιες τις ανασφάλειες, οι οποίες έχουν, τις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από το ίδιο το ρυθμιστικό πλαίσιο ε, το υφιστάμενο. Αυτά όλα θα πρέπει να τα δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν εδώ. τα οποία θέτουν κάποιες ε, ερωτήσεις. Αναφερθήκατε κύριε Ρολάν στο θέμα της ε, περιοχής, της περιφέρειας. Είμαι από μια περιοχή όπου έχουμε πολλές παλιές βιομηχανίες. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια εμπειρία περιφερειακή, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την πρόοδο, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί και σε άλλα σημεία, σε άλλε περιοχέ, όπου υπάρχει μια παλιά, για παράδειγμα, χαλιβουργία που αντιμετωπίζει προβλήματα, ε, προβλήματα τα οποία μπορούμε να τα κοιτάξουμε στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλήματα τα οποία σχετίζονται με το επίπεδο των επενδύσεων ενδεχομένω. και άλλα τέτοια προβλήματα. Έχετε κάτι τέτοιο να μας αναφέρετε για την επίλυση προβλημάτων σε ό,τι αφορά δηλαδή τις ε, τοπικές αδυναμίες και τις, ε, τα τοπικά προβλήματα ενός τόπου όπου ο κόσμος ενδεχομένω έχει την αίσθηση ότι δεν έχει ελπίδα, δεν έχει μέλλον. στο τομέα της ε, χαλιβουργίας. Όταν ε, ο κόσμος πραγματικά νιώθει ότι δεν έχει ελπίδα. Πείτε μας δύο κουβέντες για ε, τα θέματα αυτά που είπατε. Όταν σας μιλάω για 40 χρόνια ε, εμπειρία 40 χρόνων ως συνδικαλιστής. Στο νότο των Βρυξελών έχω να σας πω τεστρεοποιήθηκα ως συνδικαλιστής και το βασικό πρόβλημα είχε να κάνει ε, με επιχειρήσεις που έκαναν από τη μια μέρα στην άλλη στο Λουξεμβούργο του Βαλιγίου Και πρέπει να σας πω ότι χάρη στα ευρωπαϊκά ταμεία Χάρη λοιπόν στην κινητοποίηση των ταμείων αυτών, χάρη στην κινητοποίηση του, συνολικού, του, του συνόλου των φορέων τη περιοχή, όλη η περιοχή κινητοποιήθηκε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τέτοιου καταστάσει. Όταν λέω για, όταν μιλάω για φορεί, μιλά, μιλάω και για τι οργανώσει των ε, επιχειρήσεων, τι πολιτικέ ενώσει, τι πολιτισμικέ ενώσει, τι ενώσει των εργαζομένων. Όλοι μαζί λοιπόν καταφέραμε να ανασυνθέσουμε αυτή την περιοχή και σε ό,τι αφορά τον διασυνοριακό χαρακτήρα σε συνεργασία και με τη Γαλλία και έτσι καταφέραμε να ε, δημιουργηθούν νέες θέσεις ε, απασχόλησης, πολύ πιο καλές ποιοτικά από τις παλιές θέσεις. Αλλά, και αυτό το άλλο είναι σημαντικό, αυτοί που ξαναβρήκαν ε, θέση απασχόλησης στη συνέχεια ήταν ουσιαστικά τα παιδιά αυτών που είχαν χάσει τη δουλειά τους, γιατί η διαδικασία αυτή παίρνει χρόνο. Άρα, το πολύ σημαντικό στοιχείο που ανέφερες είναι η πρόληψη σε ό,τι αφορά το θέμα της αναδιάρθρωσης ε, να γίνεται ε, ενεργά και στην ώρα του. Εγώ είμαι από την περιοχή του Σαρλυρουά που έχουμε ζήσει πολλά δυστυχώς ε, περιστατικά που έχουν κλείσει μεγάλες επιχειρήσεις και την έχουμε γνωρίσει όλη αυτή την δυστυχία όταν έκλεισαν όλα τα ανθρακοριχεία κτλ. και όλες οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Έχουμε και την εταιρεία Caterpillar η οποία επίση έκλεισε, κλείνει σήμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν για μια περιοχή η οποία εφίσταται απανοτά σοκ να ε, και πάλι στα πόδια τη. Και αυτή η πραγματικότητα, δεν φταίει κανεί. Αλλά δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα μαύρα και άραχνα. Θα πρέπει να δοθεί ένα νέο δυναμισμό στην περιοχή αυτή, όπου εδώ και πολλέ γενιές οι προοπτικέ είναι πάντα αρνητικέ. Υπάρχουν όμω λοιπόν μέσα και εργαλεία. Η κινητοποίηση όλων των κοινωνικών φορέων με την ευρεία ε, έννοια αλλά όσο και να σα φαίνεται περίεργο, ε, έχει σημασία και ο πολιτισμικός παράγοντα και οι πολιτισμικοί φορείς. Όχι μόνο αυτοί φυσικά, θα πρέπει να κινητοποιηθούν και άλλοι παράγοντε. για να δοθεί ε, μια εικόνα ε, περηφάνεια, αν θέλετε, και για του ανθρώπου αυτού. Να μπορούν να αισθάνονται περήφανοι και αισιόδοξοι για το μέλλον του. Σε ό,τι αφορά την αντιάθραση, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει επαρκή σε πρόληψη και ενεργή δραστηριοποίηση εκ των προτέρων και να υπάρχουν και κάποιοι πυρήνε ε, μετάλλαξης ε, και μεταρρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, να οργανωθεί η συνοδεία, η καθοδήγηση των εργαζομένων από άλλους εργαζόμενους ενδεχομένως σε ό,τι αφορά την ανα διάθρωση της εργασίας τους, την ε, νέα εκπαίδευσή τους, την νέα κατάρτισή τους για νέους ορίζοντες. Και αυτό σημειώνει πολύ θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ε, κατάρτιση και την νέα αξιοποίηση των εργαζομένων αυτών στο πλαίσιο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ και σας κύριε Πρίνσκι, όπου πρέπει να πω ότι αναφερθήκατε στην αντίλατη εργασία. Και ψάχνετε λύσεις για το θέμα της αντιληπτής εργασίας και μάλιστα επί σειρά μηνών ψάχνατε λύσεις πέρσι. Κάντε μας μια σύντομη εισαγωγή. Τι μπορούμε να κάνουμε. για να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται τα επίπεδα της αντιληπτής εργασίας. Και τι εννοείται με το αντιληπτή εργασία. Well, <clears throat> to perhaps make a... Για να μην μακρηγορήσω, θα ήθελα να ξεκινήσω από το τέλος. Με συναπόφαση, λοιπόν, δημιουργήθηκε μία πλατφόρμα από το Μάρτιο ε, του φετινού έτους, λεφτή σχετική απόφαση για την αντιμετώπιση της αντίρρητης εργασίας. Τι σημαίνει λοιπόν αντιμετώπιση και πρόληψη, αλλά και α, αντιμετώπιση της αδελφής εργασίας και έβρεση τρόπων με τις οποίους μπορεί να ενταχθεί κανείς στο κανονικό σύστημα εργασίας όταν είναι στην αδελφή εργασία. Και αυτό εμπλέκει και τους ε, αντιπροσώπους και εκπροσώπους της των ευρωπαϊκών οργανισμών, των ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων και ούτω καθεξής. Και θα ήθελα να σας πω ποια ήταν τα αποτελέσματα της δεύτερης συνάντησης της πλατφόρμας. 10 Οκτωβρίου έλαβε χώρα η συνάντηση αυτή, όπου και τροποποιήθηκε το πρόγραμμα εργασίας, όπως είχε προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν πάρα πολύ φιλόδοξο και πολύ λεπτομερές το πρόγραμμα εργασίας. Έχει να κάνει με την καλύτερη κατανόηση της φύσης της τη εργασίας, πώς συλλέγουμε στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες. Και πώς καταλήγουμε και σε κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις, γιατί αυτό περιλαμβάνεται στην εντολή της ε, πλατφόρμας. Κάποια συμπεράσματα δηλαδή, σε ό,τι αφορά. Τις συστάσεις λοιπόν αυτές. Θα ήθελα να πω το εξής. Ε, ήταν πάρα πολύ σημαντική η συμβολή της Eurofound. Οι μελέτες, οι έρευνες, πολύ λεπτομερείς και μας χρησιμεύσαν πάρα πολύ και απέδειξαν ότι η αντιμετώπιση της ε, αντρέτης εργασίας έχει να κάνει και με την πρόληψη αυτής. και τη ρύθμιση, τη διευθέτηση των περιπτώσεων αυτών από τα συνδικάτα, από τις εταιρείε έχει προκύψει ότι είναι πραγματικά όλοι εντυπωσιασμένοι από τη δέσμευση και τον ανεργό τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί την πλατφόρμα. Η κυρία Ουλσκοκ ε, μας ε, είπε ότι πρέπει να κατανοήσουμε την ε, αδηλωτή εργασία και στους ε, τρεμερείς διαλόγους και στο κοινοβούλιο πρέπει να σας πούμε ότι υπήρχε η αίσθηση ότι ο, ο όρος αυτός υπάρχει από την ε, δεκαετία του 90 και τι ορίζεται ότι η αδελφή εργασία δεν είναι μαύρη εργασία, δεν είναι παράνομη, απλά δεν δηλώνεται όπως θα έπρεπε. από πλευρά φορολογική, εργασιακών δικαιωμάτων κτλ. Αλλά προκύπτει ότι η έννοια της αντιλήτης εργασίας και η τρέχουσα διαμόρφωση και πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αδήλωτη εργασία είναι πάρα πολύ περίπλοκη και είναι πολλές οι περιοχές και μεταξύ της ε, τη της εργασία, εργασίας, της εργασία εργασίας κτλ. Και πιστεύω ότι η πλατφόρμα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν πολλά θέματα που συζητήθηκαν σήμερα το πρωί σε ό,τι αφορά την ποιότητα της εργασίας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, και νομίζω ότι έτσι γνωρίζουμε πολύ περισσότερο το τι περιλαμβάνει η εργασία. Ο κ. Γκαρνιέ τώρα, ο κ. Γκαρνιέ, ο οποίο είναι γενικό γραμματέα της Γαλλικής Ομοσπονδίας Εργασίας και Άντι Νέρινερ, σύμβουλος σε υπουργικό επίπεδο στο Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Απασχόληση τη Φιλανδίας. Κύριε Γκαρνιέ, να ξεκινήσω με εσάς. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το πλαίσιο, τη συμφωνία πλαίσιο μάλλον, το οποίο διαπραγματεύτηκαν οι κοινωνικοί εταίροι για την ποιότητα της εργασίας και την ισότητα των φύλων. Λειτουργεί. Τι μαθήματα μπορούμε να πάρουμε από αυτήν. Είναι δύσκολη αυτή η συμφωνία πλαίσιο στην εφαρμογή της, στην υλοποίησή της. Θα το συστήνετε στους συνδικαλιστές σε άλλες χώρες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις σε λίγα λεπτά. Θα χρειαζόντουσαν ώρες και ώρες. Λοιπόν, για τη συμφωνία όσον αφορά την ποιότητα ε, εργασίας στην εργασιακή ζωή. Για να το εξηγήσουμε αυτό πρέπει να πάμε λίγο πίσω στη δεκαετία του 80 και 90. Ε, στις επιχειρήσεις μιλούσαμε για συνθήκες εργασίας και ασχολιόμασταν κυρίως με τις υλικέ συνθήκες εργασίας. Την έκθεση, στην θέρμανση, σε διάφορες ουσίες και σιγά σιγά αναπτύσσονταν και νέοι κίνδυνοι, η ψυχοκοινωνική, οι συνέπειες ε, μεγάλων μερών εργασίας, η κόποση στην εργασία, η επίπονη εργασία. Αναγνωρίστηκαν δηλαδή διάφορες εκθέσεις στην εργασία που μπορεί να επηρεάσουν την καλή υγεία του εργαζόμενου. Και σε αυτή την εξέλιξη πρέπει να προσθέσουμε και την εξέλιξη στις μεθόδους management. Κάνουμε όλο και περισσότερες ε, εκθέσεις, λαμβάνουμε υπόψη μας και οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία και διαπιστώνουμε ότι χρησιμοποιούνται πιο πολύ και τα ψηφιακά. Προστίθενται το στρες, η διάκριση στους χώρους εργασίας και για να λυθούν όλα αυτά κάνουμε ένα νόμο, ο οποίος δημιουργεί μια νέα υποχρέωση για διαπραγματεύσεις στην επιχείρηση. Και τελικά φτάνουμε στα διάφορα στρώματα που μας εξήγησε και ο Ρολό λιγάκι, κάτι σαν τα λαζάνια. Και βάζουμε το ένα ζήτημα πάνω στο άλλο, σε στρωμάτωση, χωρίς όμως να βλέπουμε και τη διασύνδεση μεταξύ τους. Μία έκθεση το 2010 που δόθηκε στον τότε Πρωθυπουργό, που ονομαζόταν «Ευημερική αποτελεσματικότητα στην εργασία», οδήγησε σε συνειδητοποίηση και σε εθνικές διαπραγματεύσεις. Με συμφωνία που καταλήξαμε το 2013 που θέτει δύο ζητήματα. Το ένα είναι η ποιότητα στο χώρο εργασίας που αποτελεί μέρος της ε, γενικότερης απόδοσης της επιχείρησης. Αν δηλαδή ο εργαζόμενος κάνει μια δουλειά ποιότητας αναγνωρισμένη, τότε έχει και καλύτερες επιδόσεις. Και έπειτα υπάρχει και το θέμα της πραγματικής εργασίας, το οποίο δεν συζητιέται στη... στους κοινωνικούς διαλόγους και η συμφωνία προτείνει στις επιχειρήσεις να πειραματιστούν σε έναν άλλο τρόπο διευκρινίζοντας πιο συγκεκριμένα την πραγματικότητα που ζει ο κάθε εργαζόμενος, να αφήνουμε τον εργαζόμενο να εκφράζεται, να ξαναθέτουμε το ζήτημα της οργάνωσης εργασίας στο σύνολό της, αλλά και τονίζοντας τη συμφιλίωση της ε, ιδιωτικής ζωής με την εργασιακή. Αυτή η συμφιλίωση είναι ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να κοιτάξουμε περισσότερο σε βάθος. Αλλά η κατάσταση δεν μας το επέτρεψε να το κάνουμε με την εργοδοσία. Όταν όμως βλέπουμε τα διάφορα βαρόμετρα, τις διάφορες έρευνες για το θέμα αυτό τα τελευταία χρόνια, η προσδοκία των μισθωτών για τη συμφιλίωση αυτή προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, διαπιστώνουμε ότι έρχεται σε τρίτη θέση μετά την αναγνώριση στην εργασία και πριν από τις αμοιβέ. Άρα είναι ζήτημα για αυτού. Στη συμφωνία αυτή τίθεται και το θέμα της ισότητας στην εργασία είχε επίσης να κάνει με ένα νόμο της αποχής εκείνης και διευκόλυνε την επιστροφή στις επιχειρήσεις των γυναικών μετά από γονική άδεια. Και ακολούθησε και η γονική άδεια που περιλαμβάνονται και οι άντρες. 98,2% δεν ξέρω τώρα αν είναι άντρες ή γυναίκες. Δεν αναφέρονται όμως όλα τα θέματα που μπορεί να οδηγούν σε δυσκολίες, σε διάκριση στις επιχειρήσεις. Δεν έχουμε έναν πλήρη κατάλογο, αλλά προσπαθήσαμε να προωθήσουμε μια συστημική προσέγγιση. Γι' αυτό εξάλλου ε, απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις που διασφαλίζουν την ασφάλεια, εφόσον έχει υπάρξει συμφωνία, έτσι, από το νόμο αλλά πρέπει να έχει υπάρξει συμφωνία. Συστημική λοιπόν συμφωνία βασίζεται στο διάλογο και σε διάγνωση που γίνεται στις επιχειρήσεις και όπου συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Βασιζόμαστε στην πραγματικότητα, γιατί εκεί έχουμε τις πραγματικές ερωτήσεις. Δεν υπάρχει συνταγή θαύμα, ούτε ταμπού. Χρειάζεται χρόνος. Και εδώ είναι που υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία, δηλαδή πώς θα γίνει η αλλαγή, πώς θα αξιολογηθεί, πώς θα συνοδευτούν οι εργαζόμενοι και θα έχουν κάποια κατεύθυνση και θα είναι που χρειάζονται διάφοροι δείκτες για να αξιολογηθεί η διαδικασία αυτής της επιχειρήσης. Με ρωτήσατε αν λειτουργεί. Ε, δεν είναι απλή απάντηση. Υπάρχουν αρνητικά στοιχεία. Η οικονομική κατάσταση που επιδεινώνεται, υπάρχει ανεργία που αυξάνεται. Υπάρχουν και άλλες δυσκολίες, η, είπαμε έλλειψη σίγουρης δουλειάς, οι εύκολες απολύσεις. Έπειτα το ΕΜΕΝΤΕΦ που είναι εργοδοσία στην χώρα μας δεν επένδυσε σε τέτοια συμφωνία. Είναι οι θεσμοί, τα συνδικάτα που έχουν προχωρήσει. Έπειτα ποιότητα ζωή στην εργασία με αρχικά QVT, ξεκινάει από συζήτηση στις επιχειρήσεις. Δεν προτείνουμε διάβημα που να βασίζεται στην ε, πραγματικότητα στην εργασία, αλλά σε κάποια στερεότυπα. Και μιλάμε για την ευτυχία στην εργασία, φροντίζουμε για μαθήματα γιόγκα, για στάζ, ε, κάποια, κάποιες ε, εκδηλώσεις όπως συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι για να έχουν καλύτερε σχέσει μεταξύ του. Η επιχείρηση δηλαδή ασχολείται με τα περιφερειακά ζητήματα τη εργασία και όχι με την εργασία αυτή καθ' αυτή. Και ο άλλο κίνδυνο μέσα στα όποια θετικά για την ενίσχυση της ευτυχίας ε, στην εργασία είναι ότι αγνοούμε τις δυσκολίες των εργαζομένων. Υπάρχει ένα θέμα στάσης. Στις μεγάλες επιχειρήσεις κυρίως και λιγότερο στις μικρές είναι, λες και όλα αυτά αφορούν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τις μικρές. Όμως θα σας πω ποια είναι τα αρνητικά. Υπάρχουν και θετικά βέβαια. Η ασφάλεια σε εθνικό επίπεδο αναγνωρίζεται πλήρως. Χρειάζεται εξυγχρονισμός. Οπότε ο διάλογος με τους εργαζόμενους αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της ζωής στην επιχείρηση και ένα βασικό πυλώνα των προγραμμάτων της κυβέρνησης για την ασφάλεια και την υγιεινή στον χώρο εργασίας. Το κράτος δεσμεύεται για την υγεία στην εργασία και υπάρχει και ένας χάρτης πορείας από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που ενισχύει την ποιότητα στην εργασία. Ένα άλλο θετικό δεν έχω παράδειγμα που να δείχνει κάποια επιχείρηση η οποία έχει κάνει πίσω σε σχέση με αυτά τα ερωτηματολόγια για την ποιότητα στην εργασία. Και έχω να σας δώσω πολλά παραδείγματα. Σε μερικές επιχειρήσεις γίνονται αναδιαρθρώσεις. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι απολύονται τη στιγμή που γίνεται αναδιάρθρωση. Είναι αλήθεια. Πώς τώρα σε μια βιομηχανική ζώνη μια τέτοια διαπραγμάτευση για την ποιότητα στην εργασία οδηγεί σε προσαρμογή των ωραρίων ή επιτρέπει την δημιουργία σχέσεων ανάμεσα στη διεύθυνση και του εργαζόμενου ακριβώ για να φιλιωθεί η επαγγελματική με την προσωπική ζωή ή σε μια αυτοκινητοβιομηχανία πώς λαμβάνεται υπόψη, πώς δηλαδή εισακούονται και ανταποκρινόμαστε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι για να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους. Έχουν εντοπιστεί πάρα πολλέ δυσλειτουργίε, 80% των δυσλειτουργιών ε, αυτών οδήγησαν σε απαντήσεις που βρήκαν οι ίδιοι οι μισθωτοί. Θα μπορούσα να πολλαπλασιάσω, να σας πω πολύ περισσότερα παραδείγματα. Η προσπάθεια αυτή για την ε, βελτίωση της ποιότητας ε, ζωής στην εργασία εξαρτάται από το κατά πόσο εμείς μπορούμε να προτείνουμε κάτι διάρκειας. Στην αυτοκινητοβιομηχανία, για να επανέλθω πάλι, έχουμε περάσει το δεύτερο στάδιο. Προχωρήσαμε στο πρώτο που πέτυχε. Δοκιμάσαμε πώς σε όλους τους χώρους της επιχείρησης θα γενικευθεί το παράδειγμα που πέτυχε σε ένα χώρο. Οπότε όταν με ρωτάτε αν λειτουργεί, ναι λειτουργεί, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα έχουν κερδιθεί. Είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοια συμφωνία. Βεβαίω. Γιατί είναι κάτι καινούριο και όλα τα συμβούλια επιχειρήσεων είναι επιφυλικτικά. Και έρχομαι από μια χώρα που ξέρει από αυτά. Υπάρχουν προϋποθέσεις. Πρέπει το top management να δεσμευτεί. Μια τέτοια συμφωνία για την ποιότητα ζωής ε, στην εργασία είναι ένα σχέδιο που δίνει λόγο στους εργαζόμενους και οι εργαζόμενοι πρέπει να τον πάρουν το λόγο και να πούνε πράγματα. Ε, δημιουργεί προσδοκίες και πρέπει να στεκόμαστε στο ύψος των προσδοκιών. Κάπου, σε μια γαλλική επιχείρηση που κάνει λάστιχα, ελαστικά, ο, το αφεντικό είδε το αποτέλεσμα του βαρομέτρου για την ποιότητα ζωής ε, στην εργασία, στην επιχείρησή του και έκανε τα πάντα. Και είπε ότι θα έχουμε πρόβλημα αν συνεχίσουμε έτσι. Σήμερα λοιπόν σκέφτονται μια οργάνωση της εργασίας με περισσότερη συμμετοχή και ευθύνη από πλευρά των εργαζομένων. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι πώς συνοδεύουμε τις ομάδες. Και εδώ θέλουμε διαπραγμάτευση της μεθοδολογίας και μέσα για να πετύχει η διάγνωση, η παρακολούθηση και αξιολόγηση. Για το χειρότερο κίνδυνος στην κοινωνία μας είναι η δικτατορία του τώρα πρέπει να γίνει. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία για την ποιότητα ζωή ε, στην εργασία, ε, δεν σημαίνει ότι εδώ και τώρα θα γίνει. Χρειάζεται χρόνος. Και η τρίτη προϋπόθεση είναι να υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αποσταθεροποιητικό από το να γίνει μια διάγνωση βασιζόμενη στην έκφραση των εργαζομένων πρέπει να ξέρουμε ότι δεν θα λυθούν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν πρέπει να μπαίνει σε αμφισβήτηση ούτε η εργοδοσία, ούτε οι εργαζόμενοι αν τα πράγματα δεν προχωράνε γρήγορα. Πολλά συνδικάτα έχουν επενδύσει σε τέτοιου είδους συμφωνίες για τις ηθίκες εργασίας, αλλά υπάρχει και επιφύλαξη, γιατί το δικαίωμα στην έκφραση των εργαζομένων δεν φτάνει. Πρέπει να ξέρουν ποιες είναι οι ανάγκες τους. Τέλος. Δεν μπορώ να τα πω σίγουρα, αλλά είμαι σε μια οργάνωση που έχουμε καταλάβει ότι δεν μπορεί να επιβάλλει ο ένα το μοντέλο του στον άλλον. Αυτό το λέω για το κατά πόσο μπορούν άλλοι να αντιγράψουν το δικό μα παράδειγμα. Η αυτοκινητοβιομηχανία στην οποία αναφέρθηκα σκέφτεται να γενικεύσει τη μέθοδο αυτή σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί όχι. Αλλά τίθεται το ζήτημα της τοπικής νομοθεσίας και της νοοτροπίας της τοπικής. Πράγματι και το ενδιαφέρον του μοντέλου αυτού για την ποιότητα ζωής στην εργασία είναι μία έννοια αρκετά ευρεία που μπορεί να προσαρμοστεί παντού. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε να πούμε. Δηλαδή η εργασία να συνδυαστεί με τις κοινωνικές προδιαγραφές, γιατί έτσι έχουμε όλοι να κερδίσουμε. Αλλιώς θα κερδίσουν οι λαϊκισμοί. Η εργασία είναι βασικό στοιχείο για την αναγνώριση των ανθρώπων και για την καλή τους συνύπαρξη. Ιδίως μέσα σε αυτή την κοινωνική και κοινωνικού τύπου κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νάρινεν τώρα. Η Φιλανδία έχει θέσει ως στόχο να είναι η καλύτερη χώρα όσον αφορά τη ποιότητα ζωής στην εργασία μέχρι το 2020. Πολύ μας αρέσουν μας κάτι τέτοια εδώ στην Επιτροπή μας. Σίγουρα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για όλους μας να σας ακούσουμε. Πείτε μας λοιπόν γι' αυτό. Τι μαθήματα έχουμε να μάθουμε, λειτουργεί αυτό το σύστημα, τι μπορούμε να μεταφέρουμε σε άλλες χώρες. Μπορεί να είναι παράδειγμα με δύο λόγια για άλλες χώρες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, όπως ξέρετε, εμείς είμαστε ε, μετριόφρονες ε, στην Φιλανδία. Πρέπει να πω ότι ένας από τους λόγους ε, ε, που ε, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε ε, με το θέμα αυτό είναι ότι έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία και επομένως μπορούμε να παρακολουθούμε τις μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Ε, λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ελπίζω ότι ε, δεν θα πω πολύ περίεργα πράγματα, αλλά δεν θα, δεν θα είναι δηλαδή πολύ υψηπετής ο λόγος μου, αλλά ούτε και πολύ ε, χαμηλός και ελπίζω ότι δεν θα σας κάνω να αναπολύετε την ώρα του μεσημεριανού φαγητού. Ε, στην ουσία εγώ θα ασχοληθώ με τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα πω πολύ θετικά πράγματα για την Eurofound. Μετά θα περιγράψω ε, το ε, ε, φιλανδικό παράδειγμα και αυτό το πρόγραμμα για το 2020 και θα αναπτύξω την ανάγκη, θα περιγράψω την ανάγκη ύπαρξης συγκριτικών στοιχείων για την έρευνα. Βέβαια πολλά πράγματα από αυτά που θέλω να πω έχουν ήδη θυγεί και από το πάνελ και θα είναι κατά κάποιο τρόπο η αντίδρασή μου σε αυτά που είπε το πάνελ. Λοιπόν, το παράδειγμα της ε, Φιλανδίας λέγεται Project Working Life 2020. Βασίζεται στην ε, στρατηγική που ξεκίνησε το 2012 και αφορά ε, την, ε, τον εργασιακό βίο. Η παρούσα κυβέρνηση ξεκίνησε με την προηγούμενη κυβέρνηση. Ε, εν τω μεταξύ άλλαξε η κυβέρνηση και άλλαξε και η σύνθεση των ε, κομμάτων. Παρόλα αυτά η δέσμευση συνεχίστηκε. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς περί τα εργασιακά στην Φιλανδία έχουν συνεχίσει με την ίδια δέσμευση η μοναδικότητα αυτού του Εβραίους προγράμματος ε, είναι ακριβώς, έγκυται ακριβώς το γεγονός ότι είναι ένα ευρύ πρόγραμμα και περιλαμβάνει από το, τα Υπουργεία μέχρι τα Ιστιτούτα ε, Ινστιτούτα Έρευνας, μέχρι τους εργαζόμενους, μέχρι ε, τους εκπροσώπους, συνδικαλιστικούς φορείς ε, κλπ. Επομένως, μέσω του προγράμματος παρέχεται μία πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών. Ε, επίσης ε, εκεί αναφέρονται ας πούμε όλα τα στοιχεία ή αλλαγές που θα ε, χρειάζονταν σε μία θέση εργασίας. Επίσης ε, έχουμε ε, ε, χρηματοδότηση για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος της εργασιακής ζωής και εμείς αντλούμε επίσης χρηματοδότηση για το στόχο αυτό και από το Κοινωνικό Ταμείο της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν κάποια κεντρικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με το πόσο δουλεύουμε στη Φιλανδία, ε, με κάποια ιδεολογικά στοιχεία ε, και με τα οποία μας οδηγούν ε, στην ανάπτυξη κάποιων στοιχείων στη θέση εργασίας και εδώ θα πω ότι ήδη ο David Βόλτεν έχει αναπτύξει το, το θέμα αυτό. Επίσης, θεωρούμε ε, και επιβεβαιώνεται αυτό από την μελέτη που μόλις ε, παρουσιάστηκε ότι η ευζοία συνδέεται άμεσα ε, με την ποιοτική θέση εργασίας. Για και βεβαίως για αυτούς τους λόγους ενδιαφέρεται και η εργοδοσία να αυξήσει την, ε, ε, την ε, ευεξία των εργαζομένων στη θέση εργασίας έτσι ώστε και η αποδοτικότητά τους να είναι μεγαλύτερη. Όσον αφορά τώρα τις διασυνδέσεις, προστασία, εργασιακές συνθήκες κλπ. Βεβαίως υπάρχει παρακολούθηση όλων των στοιχείων αυτών ε, στο project για την εργασιακή ζωή. Ε, αντλούμε στοιχεία και από την ε, Eurofound ε, όπως ε, ε, είπαμε και σας είπα και προηγουμένως, πρόκειται για έναν εθνικό στόχο. Μας ενδιαφέρουν επομένως πολύ τα εθνικά στοιχεία, αλλά μας ενδιαφέρει και να διασυνδέσουμε τα στοιχεία αυτά τα εθνικά με τις χώρες, με τα στοιχεία που αφορούν τις άλλες χώρες. Επίσης, μας ενδιαφέρει να κάνουμε αμοιβαία αξιολόγηση να δούμε σε περιφερειακό, τομεακό επίπεδο πώς λειτουργούν ε, τα πράγματα. Όλα τα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν ε, υπόψη. Να, ας πούμε, βλέπουμε ε, τα, τους διάφορους δείκτες που χρησιμοποίησε η Eurofound. Λοιπόν, όσον αφορά την ε, ε, διαχείριση ε, και την ικανοποίηση της διαχείρισης των προβλημάτων στη δουλειά, ε, βλέπουμε ότι ο μέσος όρος ας πούμε στην Ευρώπη μπορεί να, είναι 68, ε, από 68 μέχρι 83. Ε, στην Φιλανδία είμαστε στο 74% άρα πρέπει να το δούμε. Αν δει κανείς τον δίκτυ για την εντατικοποίηση της δουλειάς και την ένταση στους χώρους εργασίας βλέπουμε ότι και εμείς βρισκόμαστε περίπου στο μέσο όρο της Ευρώπης όμως ε, οι διαφοροποιήσεις ε, είναι πάρα πολύ μεγάλες αν, ε, μεταξύ των διαφόρων κλάδων και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η αλλαγή των συνθήκων εργασίας που είναι και το θέμα της σημερινής διάσκεψης. Εμείς έχουμε στοιχεία και για το θέμα αυτό προκύπτουν βεβαίως κάποια ερωτήματα. Αλλάζει η εργασιακή ζωή. Εάν η απάντηση είναι θετική, αυτές ε, οι αλλαγές αφορούν μόνο τον χώρο εργασίας ή διασυνδέονται και με κοινωνικές αλλαγές. Ε, επίσης η διασύνδεση είναι με θετικό ή με αρνητικό πρόσημο. Επίσης άλλη ερώτηση προσαρμοζόμαστε καλά στις αλλαγές ή μήπως θα ήταν καλύτερα να προλαβαίνουμε τις αλλαγές αυτές. Θα ξεκινήσω τώρα με τα τελικά μου συμπεράσματα και θα σας πω τα εξής. Πρώτον, νομίζω ότι οι εργασιακές συνθήκες παίζουν πράγματι σημαντικό ε, ρόλο έτσι ώστε να διαμορφώσουν ε, τις ε, οργανωτικές συνθήκες. Δεύτερον, σε κάθε έρευνα θα πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο, της διαφορετικές οργανώσεις, τις διαφορετικές οργανώσεις εργασίας, τις διαφορετικές νοοτροπίες, Τρίτον, υπάρχει οπωσδήποτε μεγάλο περιθώριο βελτίωσης των πρακτικών ε, ε, που ταυτοχρόνως θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας και της ε, επιδόσεως στις επιχειρήσεις. Όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν τέτοιες πρακτικές γιατί είναι προς το καλό τους. Με όλα αυτά λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερη ε, βιωσιμότητα και ε, σωστή, σωστές συνθήκες ε, εργασίας και να εγγραφούν λοιπόν αυτές οι αλλαγές στο χρονολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θέλει κανείς να υποβάλει ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες που έχουμε εδώ, γιατί έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Στο... Σας ευχαριστώ. Δύο ερωτήσει έχω να κάνω. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια ερώτηση. Προς εσάς κύρια. Είναι δεδομένο ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, έχουμε ακόμα υψηλή ενεργία, αλλά και αλλού. Εγώ είμαι η Ελίζα είμαι από την Ισπανία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, στο πλαίσιο του κοινωνικού πυλώνα, αυτό που λέγεται για τις ενεργές πολιτικές, για την ε, αγορά εργασίας και πώς ε, προσαρμόζονται σε ό,τι αφορά τη μετάβαση από την μη απασχόληση στην ενεργεία στην απασχόληση στην απασχόληση καλής ποιότητας. 64% ε, των ε, θέσεων απασχόλησης στην Ισπανία υπολογίζονται ότι είναι χαμηλής ποιότητας. Ποιες είναι λοιπόν οι προσδοκίες και πώς ε, εξασφαλίζουμε ότι ο κόσμος που βρίσκει μία θέση εργασίας από την ανεργία όχι μόνο βρίσκεται θέση απασχόληση, αλλά βρίσκει μια θέση απασχόληση υψηλή ποιότητα. Κάτι άλλο τώρα για του κοινωνικού εταίρου. Σε ό,τι αφορά και το πολιτικό μήνυμα που απέφτεινε στην αρχή η κυρία Πρόεδρο. Σκεπτόμενοι και αυτά που έγιναν στις ΕΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τεράστια διάκριση, αν θέλετε, και στα γραφήματα. Βλέπουμε ότι πάνω από το ίμιση των θέσεων απασχόληση, δεν είναι καλέ. Τι κάνουμε λοιπόν. Οι κοινωνικοί εταίροι, οι συνδικαλιστές, τα συνδικάτα, τι σκοπεύουν να κάνουν για να καταργηθούν αυτοί οι τεράστιοι διαχωρισμοί στην αγορά εργασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σερβό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε. Ναι, και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε. Αν μου επιτρέπετε καταρχάς να αδράξω την ευκαιρία για να υπογραμμίσω και πάλι την έκθεση της ανάπτυξης, την οποία την έθιξε και ο κ. Πυρίνσκι. Ας είμαστε και λίγο θετικοί. Δεν συμβαίνουν πάντα αυτά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά στέλνει τόσο θετικά μηνύματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απασχόληση. Το ποσοστό ανεργίας έχει πέσει στο 8,5% τον Σεπτέμβριο 2016 θετική εξέλιξη. Το χαμηλότερο, δυνατό, το χαμηλότερο επίπεδο που έχουμε φτάσει από το 2009, από την αρχή της κρίσης. Δεν λέμε ότι είναι θετικό αυτό, αλλά είναι μια μικρή βελτίωση που επηρεάζει όλα τα κράτη-μέλη. Εκ παραλλήλου, έχετε δίκιο. Οι θέσεις απασχόλησης που προσφέρονται δεν είναι της καλής ποιότητας πάντα. Αλλά Όντως βλέπουμε ότι οι θέσεις που δίδονται είναι όντως σε πρώτη φάση βράχοι πρόθεσμες και κακοπληρωμένες δουλειές, αλλά βλέπουμε ότι αυξάνονται και οι ποιοτικέ θέσει απασχόληση τώρα. Και θα έλεγα ότι η δυσκολία είναι ότι αυτές οι μόνιμες θέσεις απασχόλησης ε, προσφέρονται σε υψηλότερο επίπεδο εξειδικεύσης που προϋποθέτει κάποια α, εξειδικεύση, κατάρτιση, εκπαίδευση. Και νομίζω ότι αυτό ήθελα να πείτε. Εδώ λοιπόν περιμένουμε να αλλάξουν πολλά. Και ένα παράδειγμα να σας δώσω, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο με ενοχλεί στην Ισπανία. Έχετε εξαιρετικά σχολεία και κρατικές σχολές για νοσοκόμες κάθε χρόνο. Ε, βγαίνουν πολλές καλές ε, νοσοκόμες. Και τι κάνουν λοιπόν οι νοσοκόμες όπου υπάρχει ανεργία. Έρχονται στη χώρα μου που υπάρχει έλλειψη νοσοκόμων. Και χρειαζόμαστε νοσοκόμες. Αλλά αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι άδικο γιατί η Ισπανία φέρει το βάρος της εκπαίδευσης των ανθρώπων αυτών και εμείς ωφελούμαστε. Αυτό σας το λέω για να καταλάβετε πόσο μπορεί να υπάρχουν και έμεσες συνέπειες. Ο κύριος Χρυσαντίνη. Α, ή όχι. Πρώτα πρόσωπο, η εκπρόσωπος της Business Europe τότε. Ευχαριστώ. Θέλω να αντιδράσω κάπως γρήγορα σε αυτό που είπατε εσείς ότι είναι έτσι, αλλά στις χώρες, τις νέες μέλη, είναι πιο οξύο το ζήτημα. Έχουν καλά πανεπιστήμια, έχουν εξαίρετους γιατρούς κτλ. Οι οποίοι όμως μετά τι κάνουν, φεύγουν από τη χώρα και πάνε αλλού. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόκληση για την ενιαία αγορά και για την αποδοχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για το δεύτερο που είπατε, όσον αφορά τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας, δεν ξέρω σε τι διάκριση αναφέρεστε. Υπάρχει επαγγελματική στις βόρειες χώρες, όπου οι γυναίκες αναλαμβάνουν όλες τις διοικητικές θέσεις απασχόλησης και οι άντρες τις πιο ε, βιομηχανικές. Εσείς, εγώ μιλάω για μια νέα μορφή. Ανάμεσα στις ε, θέσεις απασχόλησης ε, υψηλών προσόντων και τις χειρονεκτικές. Αν δείτε τα ποσοστά που μας έδωσε η Eurofound, πάνω από τις μισθές θέσεις απασχόλησης χαρακτηρίζονται ως μη τόσο καλές. στη βιομηχανία είναι υποπίεση, είναι χαμηλής ποιότητας, που δεν έχει κανείς προοπτική σταδιοδρομίας. Απλώς και μόνο δηλαδή, κοιτώντα τα αποτελέσματα. Οι μισές θέσει απασχόλησης στην Ευρώπη φαίνεται ότι δεν είναι καλές θέσεις απασχόλησης. Πρέπει να δούμε και τα στοιχεία αλλά και την ερμηνεία. Εγώ δεν θα συμφωνούσα με τη δική σας ερμηνεία. Έπειτα, όπως και Μισελ νομίζω ότι εσείς το είπατε. Άμα δούμε το είδο σύμβαση εργασίας, στη Γερμανία για παράδειγμα, πολλοί μακροχρόνιοι άνεργοι επιστρέφουν στην αγορά εργασίας και έχουν μια σταθερή σχέση μέσα από ένα γραφείο ευρέσεως εργασίας, το οποίο ξέρω ότι εσείς το θεωρείτε επισφαλή εργασία. Ενώ στη Γερμανία καθέλω παρέτσι είναι. Γιατί είσαστε ένας εργοδότης αν έχετε τέτοια υπηρεσία βρέσεως εργασίας. Το άλλο, τι εννοούμε λέγοντας προοπτική. Εννοείται, δεν πρόκειται όλοι να γίνουν top manager, ούτε top μηχανική, δεν υπάρχουν τόσο πολλές θέσεις στην κορυφή για να μπορέσουμε όλοι να φτάσουμε εκεί. Αλλά συγχρόνως υπάρχει θέμα προσόντων, ικανότητας να αποκτήσει τα προσόντα. Γιατί μην ξεχνάμε, δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες ικανότητες και το έχουμε δει. Εσεί λέτε ότι υπάρχει αναντιστοιχία, ότι υπάρχουν τόσε θέσει απασχόληση για μηχανικού, πληροφορική κτλ. Πώ θα πάει κάποιος που έχει κάνει χειρονακτική εργασία για χρόνια και θα γίνει ξαφνικά τέτοιο ειδικό. Ε, είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί για μερικού να γίνει, αλλά για του περισσότερου δεν θα γίνει. Έπειτα, υπάρχουν και ένα σωρό δουλειέ που δεν θέλει κανεί να κάνει. Από τη χειρονακτική την παραγωγή που θεωρείται πιο δύσκολη, πιο κοπιαστική. Τώρα που έχουμε μηχανήματα, έχουμε απαλλαγή από πολλές τέτοιες θέσεις απασχόλησης, γιατί τα κάνουν τα μηχανήματα. Τώρα αρχίζει ο κόσμος όμως και λέει και ποιο είναι το νόημα της δουλειάς μου. Αν εγώ κάθομαι μπροστά σε ένα μηχάνημα και κάνω την ίδια κίνηση συνέχεια, τι νόημα έχει η δουλειά Αυτό ε, το έχουμε ακούσει ήδη από τη διάβρωση του χαρακτήρα το βιβλίο που είχαμε πριν από 50 χρόνια σχεδόν. Υπήρχε και το παράδειγμα των ε, φούρνων. Πολλοί φούρναρες τότε αρρώστεναν επειδή ανέπνεαν το αλεύρι. Που έφτανε στους πνευμονές τους και στη συνέχεια είχαμε αυτοματισμό στους φούρους. Οπότε οι φούροι που ζήμωναν, έκαναν το ψωμί και ανέπνεαν, τώρα πατάνε το κουμπί μιας μηχανής και το κάνει εκείνη. Έχασαν βέβαια τον έλεγχο της δουλειάς τους. Άρα η δουλειά τους, λένε, δεν έχει νόημα. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι είναι δύσκολο γιατί εξαρτάται από το τι δουλειά κάνει κανείς. Και εγώ πολλές φορές γράφω στον υπολογιστή μου και δεν γράφω πια με το χέρι, ενώ πολύ μου άρεσε όταν ήμουν πιο νέα. Και μένα με ενοχλεί αυτό. Ε, αλλάζει η φύση της δουλειάς. Από την άλλη μεριά, ε, χειρενεκτική δουλειά που ήταν πάρα πολύ σκληρή και δύσκολη, δεν χρειάζεται πια να την κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά έτσι χάνεις και το νόημα της εργασίας σου. Οδηγείσαι σε μια άλλη κατάσταση που πρέπει να εκτιμήσεις τα θετικά. Θέλω να πω ότι οι εξελίξεις είναι περίπλοκες και με την ψηφιοποίηση θα είναι ακόμα πιο περίπλοκες οι αλλαγές και οι εξελίξεις. Χάνουμε όντως τον έλεγχο. Όταν έχουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο οδηγάει μόνο του, χάνουμε τον έλεγχο. Εντάξει, το θέλουμε. Είναι ζήτημα κοινωνίας να αποφασίσει. Πάντως σίγουρα υπάρχει μια πρόκληση να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη σκληρή χειρονακτική εργασία και απ' την άλλη να δημιουργήσουμε ένα χώρο εργασίας και δουλειές που να εξακολουθούν να έχουν νόημα. Τι να γίνει, χρειάζονται. Τι θα κάνεις, θα βάλεις τι, τους μετανάστες να κάνουν τις δουλειές που δεν θέλουν οι άλλοι. Θα τις βάλουμε αυτές σε ένα χώρο να μην τις βλέπει κανείς και να νομίζει ότι δεν υπάρχουν. Μιλάμε για την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση είναι Πολύ καλό πράγμα. Μάλιστα. Πώς όμως ανακυκλώνεται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, κάποιος στην ε, Νότια Ασία κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά. Εμείς δεν τη βλέπουμε, εμείς βλέπουμε τα ανακυκλωμένα προϊόντα, αλλά δεν βλέπουμε από τη διαδικασία περνάνε και ποιος υποφέρει από αυτή τη διαδικασία. Οπότε εξαρτάται πω αντιλαμβανόμαστε τη δουλειά που κάνουμε. Είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που δεν είναι δυνατόν να το συζητήσουμε βάσει μιας έρευνας ή γενικεύοντας. Πρέπει να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Βυζαντίνη, εσείς τώρα. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Νομίζω υπάρχει ένα καλό παράδειγμα για να περιγράψουμε τι σημαίνει η διάκριση στην εργασία. Είναι τα αποτελέσματα του Brexit. Αν δείτε τη ψήφο των ανθρώπων στο δημοψήφισμα, θα δείτε ότι κυριάρχησε το Brexit στις περιφέρειες εκείνες όπου δεν υπάρχουν περισσότεροι μετανάστες, αλλά οι περιφέρειες όπου υπάρχουν τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, οι περιοχές που πλήγησαν περισσότερο από την παγκοσμιοποίηση, από τις κλιματικές αλλαγές, από την ψηφιοποίηση κλπ. Αυτό τώρα έχει να κάνει με το πώς ψήφισαν οι άνθρωποι. Αλλά έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 70% των νέων δεν πήγαν να ψηφίσουν όμως καθόλου. Και από αυτό το 70% των νέων πολλοί βρίσκονται σε επισφαλή εργασία. Και εδώ δεν ε, μιλάω κι εγώ, δεν καταδικάζω τις ε, εταιρείε ευρέσεως εργασίας. Όχι, είναι το λιγότερο αρνητικό παράδειγμα ατυπικής εργασίας. Υπάρχουν άλλες μορφές άτυπης εργασίας που δεν προέρχονται από αυτές τις ε, επιχειρήσεις ευρέσεως εργασίας. Λοιπόν, όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν χάσει τη δουλειά τους εξαιτίας αναδιάρθρωσης της επιχείρησής τους και ζουν επιδόματα και που δεν μπορούν να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας παρά μόνο αν δεχτούν πολύ χαμηλές, χαμηλού επίπεδου και επισφαλείς δουλειές. Και υπάρχουν αυτοί που ψάχνουν δουλειά για πρώτη φορά και δεν βρίσκουν παρά μόνο αν δεχτούν πολύ κακές συνθήκες αμοιβή και εργασία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μιλάμε για 60% του εργατικού δυναμικού. Δεν ισχύει το ίδιο στη Γαλλία ή τη Γερμανία η Φιλανδία προφανώς η Σουηδία, αλλά αν δείτε τα αποτελέσματα στις περιφερειακές εκλογές της Γερμανίας, π.χ., θα δείτε ότι μάλλον ένα 30% των ανθρώπων αυτών που ψήφισαν για την εναλλακτική για τη Γερμανία, κατά πάση πιθανότητα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας. Αν δείτε την Πολωνία, η Πολωνία έχει μια αντίστοιχη κατάσταση με αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου. Και δεν είναι σύμπτωση που στην Πολωνία έχετε το υψηλότερο επίπεδο επισφαλούς εργασίας και το μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την ε, ανάπτυξη των μισθών. 43% είναι αυτή η διαφορά. Πώς εξελίσσεται η παραγωγικότητα και πώς εξελίσσεται η μισθή αμοιβές δηλαδή. Τι κάνουμε. Πρώτον, πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρώτα απ' όλα και μετά και σε εθνικό επίπεδο αποτελεσματικά να δημιουργήσουμε μια στρατηγική για μια δίκαια μετατροπή στην Ευρώπη. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε δηλαδή, είτε πρόκειται για διαφορετικές αλλαγές, είτε πρόκειται για την παγκοσμιοποίηση, είτε πρόκειται για την κλιματική αλλαγή, την ψηφιοποίηση της οικονομίας. Να μην καθόμαστε και να κοιτάμε να συμβαίνει να παρακολουθούμε δηλαδή με σταυρωμένα τα χέρια. Όχι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο και θα το αντιμετωπίσουμε με τις κατάλληλες πολιτικές. Δεν μπορεί απλώς να λέμε ότι θα καταστραφούν θέσεις εργασίας αλλά θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Όχι, γιατί δεν βλέπουμε να δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Αν λοιπόν για τις 10 που καταστρέφονται μπορείτε να φτιάξετε 11 και θέλετε να φτιάξετε 11, κάτι πρέπει να κάνετε. Να εκπονήσετε τις κατάλληλε πολιτικές για να αντιμετωπίσετε τέτοιες προκλήσεις. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος Γιούνκερ στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από μερικούς μήνες. Είπε ότι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που να προστατεύει τον κόσμο, τους πολίτες, να είναι σαν καταφύγιο για αυτούς. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα κατάλληλο δίκτυ κοινωνικής προστασίας Οπότε, λαμβάνοντα υπόψη και την ευελιξία, να μπορούμε συγχρόνω να προστατεύουμε τον κόσμο, να νιώθει ασφαλή ο κόσμο μέσα στην κοινωνία. Και μόνο έτσι θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα. Και νομίζω ότι αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα που αναπτύσσει την κοινωνική πτυχή εκείνη των κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι η σωστή προσέγγιση. Πρέπει να ενισχύσουμε τον πυλόν αυτό και να διασφαλίσουμε ότι στον πυλόν αυτό θα έχουμε και συγκεκριμένε δράσει με τις οποίες να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τον κόσμο. Γιατί αν δεν τα κάνουμε για τον κόσμο, αν δεν δει αποτελέσματα συγκεκριμένα, καταλαβαίνετε ότι θα ξεπεραστούμε από τέτοιου είδους αρνητικά κύματα όπως αυτά που διαδίδονται στην Ευρώπη τελευταία. Είναι θέμα των πολιτικών, αλλά είναι θέμα και των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας συνολικά. Πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Και το τελευταίο που πρέπει να κάνουμε γιατί ωραία, ακόμα και αν έχουμε μια καλή δίκαια μετατροπή, ακόμα και αν έχουμε υψηλέ προδιαγραφές, ακόμα και αν έχουμε συστήματα κοινωνικής προστασίας που να έχουν καλές επιδόσεις, αν δεν δημιουργήσουμε νέες ε, θέσεις απασχόλησης, θα είναι μια τρύπα στο νερό. Μπορούμε να συζητάμε για τι καλύτερε συνθήκε εργασία στον κόσμο που θα εφαρμόσουμε στην Ευρώπη, αλλά αν δεν έχουμε δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τότε έχουμε πρόβλημα που δεν λύνεται. Και ο μόνος τρόπος είναι να σπρώξουμε για την οικονομική ανάκαμψη, την οικονομική ανάπτυξη. Τα δύο μέσα που έχουμε σήμερα υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης, από τη μια μεριά είναι οι επενδύσεις και έχουμε το σχέδιο Juncker, που για μας δεν φτάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι είναι. Να ενισχύσουμε τις επενδύσεις για να έχουμε ανάκαμψη της οικονομίας οι δημόσιε και ιδιωτικέ επενδύσει τα τελευταία 5-10 χρόνια στην Ευρώπη είναι μηδέν. Έχουν καταρρεύσει. Τίποτα. Τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Αν λοιπόν δεν αλλάξει αυτή η τάση προς τα κάτω, δεν θα έχουμε και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Και το άλλο, και λυπάμαι που το επαναλαμβάνω, είναι η μισθή. Ο Μισελ είπε ότι πρέπει να ενισχύσουμε και την εσωτερική ζήτηση, όχι μόνο την παραγωγικότητα. Γιατί εντάξει οι εξαγωγέ μα στην Ευρώπη, αλλά πάλι αποτελούν μικρό μέρο τη οικονομία μα. Το μεγαλύτερο μέρο τη ε, ευρωπαϊκή οικονομία είναι η εσωτερική ζήτηση, η οποία έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Καταστρέφουμε τη δυνατότητα του κόσμου να αγοράσει αγαθά, υπηρεσίε. και να αποκτήσει καλύτερες συνθήκες ε, ζωής μέσω της ενίσχυσης της εσωτερικής ζήτησης. Και αυτό είναι πρόβλημα όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και για τις επιχειρήσεις. Γιατί θα έχουμε όλο και περισσότερο από πληθωρισμό και τελμάτωση και δεν θα έχουμε ευκαιρίες για παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα για το μέλλον. Τέλος, όταν σκεφτόμαστε, όπως είπε και η Ρενάτα πριν, ανάμεσα στην παραγωγικότητα και τους ε, μισθούς, ποια θα είναι η σχέση. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και δύο ακόμα παράγοντες. Αυτή τη διαφορά που υπάρχει, πώς τη χρησιμοποιούμε. Γιατί αν είναι μόνο για τα κέρδη, τότε δεν ενισχύει την οικονομία. Αν πηγαίνει στις επενδύσεις, στην ποιότητα, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, τότε ναι, η διαφορά αυτή μεταξύ των δύο μπορεί να δημιουργήσει απασχόληση. Δυστυχώ τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη η διαφορά ανάμεσα στην παραγωγικότητα και την ε, εξέλιξη των μισθών δεν επενδύεται στην οικονομία. Πηγαίνει στα κέρδα, πηγαίνει στη γερδοσκοπία, αλλά όχι σε βελτίωση τη οικονομία. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και το άλλο είναι ότι αν η διαφορά είναι υπερβολικά μεγάλη, τότε οι ανισότητε που προέρχονται από αυτή την υπερβολικά μεγάλη διαφορά επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα, την ε, παραγωγικότητα κλπ. Και οι δαπάνες, οι δημόσιες δαπάνες δεν γίνονται με το σωστό τρόπο γιατί πρέπει να τις σταθμίσεις. Άμα δεν έχεις καλή κατάσταση δαπανάς αλλά είναι επιδόματα αυτά και δεν είναι δαπάνη με το σωστό τρόπο. Συνεπώς όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με ρεαλιστικό τρόπο. Δεν μπορούμε απλώς να λέμε ότι όλα πάνε καλύτερα. Ναι εντάξει ίσως κάτι πηγαίνει καλύτερα, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα και ο πρώτος τρόπος για να τα αντιμετωπίσουμε είναι να αναγνωρίσουμε ότι τα έχουμε και να προσπαθούμε να βρούμε μια διέξοδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σύντομη παρέμβαση από τον κύριο Ρολάν τώρα πολύ σύντομη. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι προφανώς ε, πολιτική η ερώτηση που θέτεται. Η... Το χάσμα που υπάρχει μεταξύ της επισφαλούς εργασίας ε, χαμηλής ποιότητας και των καλών θέσεων απασχόλησης που είναι υψηλής ποιότητας είναι πραγματικά ένα θέμα πολιτικό αυτό. Πρέπει να το αποφύγουμε και θεωρώ ότι έχουμε εργαλεία και μέσα στη διάθεσή μας σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε θέματα κατάρτιση και εκπαίδευση, γιατί έχουμε προβλήματα εδώ πέρα. Θα πρέπει να δοθεί αξία στα τεχνικά επαγγέλματα, τα χειρονακτικά, όπου έχουμε προβλήματα και έλλειψη ε, εργατικού δυναμικού. Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει ένα σωστό προσανατολισμό. Και υπάρχουν ε, πολλά άτομα τα οποία δεν θα έχουν ασφαλώς πολύ υψηλό επίπεδο εξειδικευσής, αλλά χρειάζεται ένα άλλο επίπεδο απασχόλησης που θα έχει την αντίστοιχη κοινωνική και οικονομική αξία. Και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας βοηθήσει προς την κατευθύνση αυτή και νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το Εράσμους, να πρέπει να υπάρχει μια σωστή εκπαίδευση σε, ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό υποστηρίζεται και από άλλε πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προ αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον. Και τώρα, συντομία, επόμενο ομιλητή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να απαντήσω σε ό,τι αφορά τα θέματα που αναφέρθηκαν για την έκθεση και τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τι θέσει απασχόληση καλή και κακή ποιότητα. Δεν θέλουμε να πούμε σε καμία περίπτωση ότι οι μισές δουλειές ε, είναι κακές. Όταν κοιτάμε τα, τις ομάδες που εκπροσωπεί η Αγνές, ουσιαστικά τι κοιτάμε. Ποιες δουλειές έχουν λίγο πολύ τέτοια χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό κάναμε την ομαδοποίηση σε πέντε κατηγορίες. Οι ομάδες αυτές παρουσιάζουν λοιπόν κάποια αντίστοιχα χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την ποιότητά του. Το 19% για παράδειγμα, το οποίο ε, χαρακτηρίζουμε ως χαμηλής ποιότητας. Ε, πραγματικά, εδώ παρατηρούνται απαντήσεις χαμηλής, ε, μάλλον απαντήσεις κακές σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που έχουμε εντοπίσει. Αλλά δεν είναι παράνομες θέσεις εργασίας ή το 13% που είναι υποπίεση, δεν σημαίνει ότι είναι ακατάλληλες στις κακής ποιότητας, απλά έχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Η ομάδα λοιπόν χαμηλής ποιότητας παρουσιάζει λίγο τρευνοϊκά στοιχεία σε όλες τις διαστάσεις και θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Δύο άλλες παρατηρήσεις, επιτρέψτε μου, για το κατά πόσο το ποτήρι είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Και εδώ θα ήθελα να πω δύο συγκεκριμένα πράγματα. Στην έκθεση συζητάμε ένα από τα σημαντικά ζητήματα για την ασφάλεια και την υγεία, κατά πόσον είναι σωστά ενημερωμένοι οι εργαζόμενοι για την ασφάλεια και την υγεία στην αγορά εργασία, στον χώρο εργασία, Είναι θετικό το αποτέλεσμα. Στη μεγάλη πλειονότητά του είναι καλά ενημερωμένοι οι εργαζόμενοι. Πάνω από 10% ε, μάλλον ένα 10% στην Ευρώπη λέει ότι δεν είναι σωστά ενημερωμένο. Αλλά έχουμε υψηλό αριθμό των όσων είναι εκτεθειμένοι σε υψηλό κίνδυνο που δεν είναι σωστά ενημερωμένοι. Και στις μικρές επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερο το ποσοστό αυτό το μη σωστά ενημερωμένων. Επίσης, εκεί που δεν υπάρχει εκπροσώπηση των εργαζομένων, εκεί που υπάρχουν επισφαλή συμβόλαια, αλλά γενικά τα στοιχεία είναι Αλλά ο διάολος κρίνει τις λεπτομέρειες και ένα τελευταίο στοιχείο. για το ρόλο της βιώσιμης απασχόλησης και πώς μπορεί να καταστεί μια θέση απασχόληση βιώσιμη, δεδομένη και τη δημογραφική αλλαγή. Και βλέπουμε ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά, κάποιε από τι συνθήκε τη εργασία, βλέπουμε ότι υπάρχει σε κάποιε περιπτώσει ε, μετάβαση σε νυχτερινή εργασία, ε, υπάρχουν ε, προβλήματα κοινωνικά, εργασιακά Εκεί προφανώ ο κόσμο ε, έχει πιο πολλέ πιθανότητε να αναφέρει ότι δεν σκοπεύει να συνεχίσει εργασία μετά τα 60. Και να πω ότι πολλά εξαρτώνται από τη σωστή διαχείριση τη ποιότητα, από τι τοπικέ δράσει, από τη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού, του κοινωνικού διάλογου σε τοπικό επίπεδο. Και αυτά, ξέρετε, δεν είναι πράγματα τα οποία απαραίτητα κοστίζουν πολλά χρήματα. Μπορούμε να τα εφαρμόσουμε με απλό τρόπο. Ευχαριστώ. Θέλετε να κάνετε ερώτηση, λέει η Πρόεδρος. You press the red button. Or the button, perhaps. Ανοίξτε το μικρόφωνο, λέει η Πρόεδρος. Thank you very much. University of Oxford. Σας ευχαριστώ από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Θα ήθελα να επανέλθω στα αυτά που είπε ο κύριος Πυρίνσκι, πολύ ενδιαφέροντα, ότι η έρευνα καταδεικνύει μείωση των ατόμων που θεωρούν ότι η δουλειά έχει γίνει καλά. Στη σελίδα 83 της σελίδας περιλαμβάνεται κάτι που μου κάνει εντύπωση, ότι το ίμιση των εργαζομένων θεωρεί ότι το αφορά το θέμα της ποιότητας εργασίας και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και ένα τρίτο το ποσοστό αυτό. Περίεργο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και 20 χρόνια μας λέει ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε ε, οργανώσεις ε, κατάρτισης και εκπαίδευσης για διαβίου κατάρτιση. Αλλά βλέπουμε ότι μάλλον έχουμε κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση για την κινητοποίηση της δέσμευσης και της γνώσης των ε, εργαζομένων για το όφελος, προς όφελος και της εταιρεία, αλλά και του εργαζόμενου. Ποιες είναι λοιπόν οι πολιτικές οι οποίες θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να σημειώσουμε πρόοδο στο σημαντικό αυτό θέμα. Η Πρόεδρος έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας για να δούμε κατά πόσο να μπορούμε να σας δώσουμε μία απάντηση στα ερωτήματά σας αυτά. Ο κύριος Πρίνσκι. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, πιστεύω ότι η πιο σωστή η σύντομη απάντηση είναι ουσιαστικές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Γιατί Διαφορετικά οι εργαζόμενοι μένουν σχεδόν χωρίς ε, φωνή. Πιστεύω ότι μία από τις ε, ελλείψεις ε, της διοίκησης, ας πούμε, ακόμα και σε επίπεδο κομισιών, είναι ε, που ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές ε, ε, διαπραγματεύσεις έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια και η βαθμία. Ίσως τα τελευταία δύο χρόνια η Κομισιόν έχει ξανά ξεκινήσει να δίνει, αρχίσει να δίνει μεγάλη σημασία στον κοινωνικό διάλογο. Έχω πάντως την αίσθηση ότι ένα μεγάλο τμήμα του κοινωνικού διαλόγου σημαίνει να ξαναμάθουμε να μιλάμε μεταξύ μας, να μιλάει ο ένας τον άλλον και βεβαίως η συζήτηση θα πρέπει να είναι ουσιαστική και ε, ε, ε ουσιώδης λοιπόν την όλη διαδικασία η οποία ξεκίνησε ε, μετά τον Μάρτιο και το Κοινοβούλιο μέσω και της δικής μας Επιτροπής Κοινωνικών ε, Υποθέσεων συνδράμει μέσω ψηφίσματος το οποίο προετοιμάζεται ε, και στο οποίο λέμε ότι ο κοινωνικός πυλώνας, εάν θέλουμε να είναι λειτουργικός, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει και κανονιστικό χαρακτήρα, θα πρέπει να διαθέτει θεσμικούς μηχανισμούς, αλλά και να διαθέτει και πόρους. Δηλαδή θα πρέπει ναι να έχει κάποιες ιδέες, αλλά οπωσδήποτε να διαθέτει και τα μέσα έτσι ώστε να υλοποιήσει τις ιδέες. Ο κύριος Σερβόσα ε, επανήλθε ε, στις ημερομηνίε ε, και στα δεδομένα, συγγνώμη, και στα δεδομένα, αλλά τα δεδομένα υπάρχουν, δεν αμφισβητούνται. Το ερώτημα το οποίο έδεσα εγώ αφορούσε περισσότερο την ε, συνέχιση του ε, υποδείγματος της σταθερότητας που είναι συνδεδεμένη με την ε, ανάπτυξη. Ο κ. Σερβός γνωρίζει βεβαίως <coughs> πολύ καλά πόσο το κοινωνικό ταμείο ε, χρειάζεται πόρους ε, το Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης έτσι ώστε να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, έτσι ώστε να προωθήσει τα κοινωνικά στοιχεία της οικονομίας Ε, μέχρι τώρα η Κομισιόν ήταν πιο δογματική, ε, έβαλε λίγο νερό στο κρασί της μετά από τις εμπειρίες της Πορτογαλίας, της Ισπανίας κλπ. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί μια πιο ισχυρή πολιτική έτσι ώστε να αλλάξουν οι τάσεις, να υπάρξει ανάκαμψη, να ε, ξεπεραστεί και αυτή ε, η αποτελμάτωση των μισθών και των αμοιβών. και νομίζω ότι δεν θα πρέπει απλώς ε, να κάνουμε έτσι μια φιλοσοφική αναγνώριση των προβλημάτων, α, θα πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να ανατρέψουμε αυτές τις διαδικασίες που οδήγησαν στον Brexit. Thank you. I'll give the floor to you in glasses over there. Thank you. Um, σας ευχαριστώ. Από το Πανεπιστήμιο του Cambridge ε, είμαι και θα ήθελα να σας κάνω την εξή ερώτηση. Να σας ευχαριστήσω καταρχάς την ε, ομάδα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος που έκανε την ανάλυση των στοιχείων και έγραψε την έκθεση αυτή. Πραγματικά εξαιρετική. Και νομίζω ότι αυτό που διαφοροποιεί από τα άλλα έγγραφα που περιγράφουν την ε, εργασία των ανθρώπων είναι ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο που αποτυπώνει τη συνθε... την πολυσυνθετότητα, την περιπλοκότητα της εργασιακής ζωής με ακριβή τρόπο, αλλά ότι αποτελεί και ένα εργαλείο επικοινωνίας με τους μη ειδικού. Ο κοινό πολίτης νομίζω ότι καταλαβαίνει ποια είναι η ώρα εργασίας. οι κατηγορίε ε, που περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή χωρί υπερβολικό επίπεδο λεπτομέρεια και υπερβολική εξειδίκευση. Είναι σημαντικό αυτό για την κατανόηση των στοιχείων. Και ο λόγο για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό αυτό, είναι τόσο σημαντικό αυτό είναι γιατί μα δίνει νέε δυνατότητε να σκεφτούμε το πώ μπορούμε ενδεχομένω να επηρεάσουμε την πολιτική μέσα από το ενεργασία αυτή. Πώ μπορούμε να, να κάνουμε κάτι το οποίο θα σημαίνει την αλλαγή. Για παράδειγμα, από την Φιλανδία μα είπε ο εκπρόσωπο ότι θέλει να προωθήσει την ε, καλύτερη ποιότητα ε, εργασία στη Φιλανδία μέχρι το 2020. Μιλάμε για ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών, μιλάμε για ανταγωνισμό μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων. Οι τομεί, για παράδειγμα, οι οποίοι δεν μπορούν ε, να συγκεντρώσουν ε, αρκετούς εργαζόμενους και σημειώνουν προβλήματα. Πώς συμπεριφέρονται Μήπως και οι εργοδότες θα πάρουν τα πράγματα στο πιο, πιο σοβαρά, χρησιμοποιώντας και τα εργαλεία που μας δίνει η έκθεση και έτσι θα μπορέσουν να προσμετρήσουν το που βρίσκονται σε σχέση με άλλες εταιρείε, σε σχέση με άλλους κλάδους και έτσι καταβάλω μία προσπάθεια για να προσελκύσουν τους καλύτερους εργαζομένους. Πώς πιστεύετε λοιπόν ότι η έκθεση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταφύσουμε καλύτερη πολιτική, με νέους τρόπους ή πρόεδρος. Θέλετε να κάνετε και εσείς μια ερώτηση για να ακούσουμε μετά τις απαντήσεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ επίσης ε, θεωρώ ότι είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Η έκθεση σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. να σας πω πού είναι ο πυρήνας της ερώτησης. Ο κ. Βιδάν είπε εισαγωγικά στην παρουσίαση του ότι διαπιστώνει μια γενικότερη επιδείνωση της ποιότητας εργασίας σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτά που είδα στην παρουσίαση, δεν έχω διαβάσει την έκθεση, αλλά Στη διαφάνεια υπερθυμών 4 βλέπουμε την ποιότητα εργασίας με την πάρδο του χρόνου και συν... κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ 2015 με το 2010 διαπιστώνουμε ότι όλοι οι δείκτες έχουν παραμένει στο ίδιο επίπεδο από το 2015, από το 2010 μέχρι το 2015 ή έχουν επιδεινωθεί, όπως η ένταση εργασίας, η οποία έχει σημειώσει ελαφριά επιδείνωση. Η μοναδική που έχει βελτιωθεί είναι η ομάδα ικανοτήτων. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Στη σελίδα 7, κοιτάξτε, στο skills and discretions της προσόντα αυτά. Βλέπουμε την ε, εκπαίδευση που ζητείτε ή δίδεται στους ε, εργαζόμενου. Εδώ υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια βέβαια. Δεν φαίνεται στη διαφάνεια κατά πόσον η ανομοιογένεια αυτή ε, σημειώνεται σε όλες τις θέσεις απασχόλησης και σε όλους τους τύπους εργασίας. Φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. μπορεί να φαίνεται, μάλλον φαίνεται ότι έχουν επιδεινωθεί σημαντικά οι συνθήκε εργασίας. Δεν έχω δει τα μακροδεδομένα, αλλά αυτό που θα ήθελα να συμπεριληφθεί, πιστεύω, θα είναι ενδιαφέρον, είναι δύο πράγματα. Προκειμένου να αξιολογήσουμε πιο καλά το πόσο έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες από το 2010. Ίσως περιλαμβάνεται στην έκθεση. Θα πρέπει να ξέρουμε όμως το καθεστώς απασχόλησης, αυτό που αναφέρεται ως καθεστώς απασχόλησης. Αυτό που θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν, δεν ξέρω αν τα έχετε τα στοιχεία αυτά, αλλά αυτό που θέλουμε να ξέρουμε είναι τι ποσοστό των αυτοπασχολόμενων σήμερα το 2015 προέρχονται από μια κατάσταση όπου ήταν μισθωτή πριν από 50 χρόνια. Ήταν δηλαδή παλιά μισθωτή και τώρα πλέον δεν είναι μισθωτή. είναι αυτοαπασχολούμενη. Ή κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε προς τα πού κινούνται τα πράγματα στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος να ολοκληρώσω. Πολύ, πολύ γρήγορα, αν θέλετε, λέει η Πρόεδρος. Μάλιστα. Τώρα στην άλλη ωραία διαφάνεια, την οποία τη βλέπουμε και τη σχολίασαν και άλλα άτομα για τα προφίλ θέσεων απασχόλησης. Κοιτάμε τις δύο χαμηλότερες κατηγορίες, υποπίεση και φτωχής ποιότητος. Αυτές οι δύο κατηγορίες. Οι χειρονάκτε είναι στις, κατηγορίε κατηγορίες αυτές. Και πάλι θα θέλαμε να ξέρουμε πώ έχουν εξελιχθεί τα πράγματα με την παράδοση του χρόνου. Σας ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση πριν το μεσημερινό διάλειμμα, λέει η Πρόεδρος, γιατί θα έχουμε και ευκαιρίε και αργότερα να κάνουμε ερωτήσει. Τελευταία ερώτηση, αν θέλετε. Πάρτε το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι από τη Δανία, που θεωρείται η πιο ευτυχισμένη χώρα, στην Ευρώπη τουλάχιστον. Έχω δουλέψει στην ασφάλεια και την υγιεινή ως ε, γιατρός, ε, στους χώρους εργασίες, όλη μου τη ζωή. Και πράγματι και στη Δανία υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το είδος της απασχόλησης και τον κλάδο της απασχόλησης. Όταν δουλεύει κανείς με ποιότητα εργασίας, οι διαφορές αυτές εξαφανίζονται. Αν θέλεις να βελτιώσεις την κατάσταση, πρέπει να ξέρεις ότι αν υπάρχει έκθεση στη σκόνη ή οτιδήποτε άλλο, Αυτό είναι επικίνδυνο για την υγεία. Αν δουλεύεις στις οικοδομές, σηκώνει βαριά πράγματα ε, και μάλιστα είσαι έξω όταν έχει κακό καιρό, υγρασία κτλ. Πάλι είναι επικίνδυνο. Ή άμα καθαρίζεις όλη η μέρα, εντάξει, όταν γυρνάς ε, σπίτι σου προφανώς και είσαι πολύ κουρασμένος. Αυτές οι διαφορές δεν ε, φαίνονται όταν μιλάει κανείς για την ποιότητα. Η ποιότητα της ζωής στην εργασία δεν πρέπει να μπερδεύεται με τα χημικά, με τα βαριά φορτία ή με τα βακτηρίδια μέσα στα φορτηγά. Φαίνεται ότι στην καμπίνα του οδηγού ε, υπάρχουν πολλά ε, βακτηρίδια. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε για τι πράγμα ακριβώς μιλάμε και τότε να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Και για να το αλλάξουμε πρέπει να έχουμε τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι θα πρέπει να συνομιλούν μεταξύ τους και να λύσουν τα προβλήματά τους στο χώρο της εργασίας. Αν λοιπόν είσαστε εργοδότης, πρέπει να είσαστε περήφιανος αν έχετε ένα χώρο εργασίας που προσφέρει αξιοπρεπή δουλειά στους εργαζόμενους και αν νοιάζεστε ώστε να θέλουν να δουλέψουν μαζί σας όλη τους τη ζωή. Και αν θέλετε να κρατήσετε περισσότερα χρόνια τον κόσμο στις δουλειές, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι και οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Άλλοι είναι πιο υγιείς, άλλοι υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες και αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας όταν ζητάτε να κάνουν τη δουλειά τους. Και όσο το ψάχνετε περισσότερο, τόσο περισσότερες διαφορές θα βρείτε ανάμεσα σε έναν υγιή 60 ετών και σε έναν μη υγιή 60. Συνεπώς, η ποιότητα της ζωής στην εργασία δεν είναι κάτι επίπεδο, δεν μπορείτε να το βάλετε έτσι σε ένα μέτρο και μόνο σε μια ζυγαριά. Ο κόσμος θα σας πει αν γι' αυτόν υπάρχει ποιότητα ζωής στην εργασία ή όχι. Πρόεδρος, κοντεύουμε να εξαντλήσουμε το χρόνο μας. Ας προσπαθήσουμε σύντομα να καταλήξουμε σε κάτι. Σχολιάστε παρακαλώ όλοι. Έτσι τρία λεπτό καθένας. Ξεκινάμε από τον κύριο Σελβός. Και μετά και όλοι οι υπόλοιποι στο πάνελ. Και τότε θα μπορέσουμε ίσως να επανέλθουμε σε κάποιες από τις ερωτήσεις που σας τέθηκαν και το απόγευμα. Ο κύριος Σελβός πρώτα. Παρακαλώ. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος, ναι. Μια σκέψη για τις δεξιότητες. Ο κύριος Ζωρολά νωρίτερα μίλησε για τη σημασία που έχει η επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση και οι βασικές δεξιότητες. Πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Και θέλω να πω ότι έχουμε ένα σχέδιο για την κατάρτιση και για τη μαθητεία. Και θέλουμε να φροντίσουμε αυτά τα προγράμματα να επεκταθούν πολύ σύντομα. Να μην πρόκειται μόνο για πιλωτικό πρόγραμμα, αλλά να γίνει ένα πραγματικό πρόγραμμα. Άκουσα τις παρεμβάσεις από το Cambridge και το Oxford για παράδειγμα, πολύ ενδιαφέρουσες. Αν δείτε λοιπόν τα 10 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, μόνο δύο ευρωπαϊκά βρίσκονται μεταξύ αυτών. Ακριβώς, η Oxford και το Cambridge, μέχρι τώρα. Γιατί θα έρθει η στιγμή όπου τα δύο αυτά πανεπιστήμια δεν θα θεωρούνται πια ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Εδώ δεν έρχομαι να εκφράσω μια θλίψη, τα γεγονότα είναι γεγονότα, αλλά λέω ότι όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια στην Ευρώπη πρέπει να βελτιωθούν. Γιατί αν θέλουμε να έχουμε τους καλύτερους μηχανικούς πληροφορικής, τους καλύτερους μηχανικούς γενικά, πρέπει οπωσδήποτε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να βγάζουν καλύτερους φοιτητές, οι οποίοι να μπορούν να δουλέψουν στην ελεύθερη αγορά και να ανταποκριθούν στις ανάγκες της. Ένα λεπτό μόνο κράτησε. Ήταν η σκέψη που ήθελα να σας μεταφέρω. Ευχαριστούμε. Τέλεια. Παρακαλώ κύριε Βεσεντίνη. Δύο σχόλια. Πρώτον, συμφωνώ απόλυτα με όσους από εσά λένε ότι θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί όταν συζητάμε τους μέσους όρους, αυτοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση αυτή λοιπόν που πιστεύω και εγώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θετική. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μπούμε στις λεπτομερίες της και να καταλάβουμε ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, χώρους εργασίας, κλάδους, ειδικέ συνθήκε εργασίας και να φτάσουμε στην πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε αν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε σε επαφή με τη Eurofound και να καταλάβουμε τις λεπτομέρειες, τι βρίσκεται πίσω από τα νούμερα που μας παρουσιάζει στην έκθεση, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για τους κοινωνικούς εταίρους και όχι μόνο, ώστε να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα αυτή την έκθεση. Δεύτερον, είμαι πεπισμένος ότι οι κοινωνικοί εταίροι είναι οι καταλληλότεροι φορείς της αγοράς για να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Εμείς πάντα επαναλαμβάνουμε ότι πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εργασιακές σχέσεις, ο κοινωνικός διάλογος, όλα τα επίπεδα, το ευρωπαϊκό, το εθνικό, το περιφερειακό, το τομεακό και στους χώρους εργασίας. Οι συλλογικέ συμβάσει, οι εργασιακές σχέσεις μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα με έναν τρόπο που να είναι ο κατάλληλο για το κάθε πλαίσιο και την κάθε περίπτωση. Οι κοινωνικοί εταίροι τα γνωρίζουν αυτά και μπορούν να κάνουν τη διαφορά μέσα σε ένα καλό σύστημα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών διαπραγματεύσεων. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Η κυρία Χόρνουγκ τώρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Συμφωνώ 100% με αυτά που μόλις είπε ο Λούκα, ότι δηλαδή χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Ο Ντέβιτ Φόντεν επίσης έχει δίκιο που είπε ότι πολλά από όλα αυτά που εντοπίζονται στην ε, έρευνα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαφοροποιημένο τρόπο σε εθνικό επίπεδο. Η κοινωνική εταίρη τώρα. Εδώ έχουμε μια πρόκληση και έχουμε μια πρόκληση γιατί είναι όλο και πιο δύσκολο να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Και αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα. Όλοι μιλάνε για τους εργαδότες. Ποιοι μιλάνε όμως για τους εργαζόμενους και για τις δικές τους υποχρεώσεις. Ερχόμαστε με πολύ μεγάλες προσδοκίες και υπάρχει η τάση να μην ε, δεσμευόμαστε. Οπότε πρέπει να δουλέψουμε και πάνω σε αυτό για να υπάρχει πραγματικά συλλογική δράση σε τοπικό όμω πολύ συγκεκριμένο επίπεδο για να κάνει διαφορά στον κόσμο. Και εδώ θέλω να πω και κάτι τελευταίο, μια κάποιο είδου προειδοποίηση. Η διαφοροποίηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν ο κοινωνικός πυλώνας αποτελέσει κενό γράμμα, τότε θα απογοητεύσει τις προσδοκίες που θα έχει δημιουργήσει και αυτό θα ήταν η καταστροφή. Γιατί εμείς από το ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε πράγματα τα οποία θα βελτιώσουν την πραγματικότητα και θα κάνει πράξη τα λόγια και όχι να δημιουργηθούν ε, έτσι κενές υποσχέσεις που δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Θέλουμε λοιπόν ο κοινωνικός πυλώνας να αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί στην πράξη να βοηθήσει τον κόσμο να βοηθηθεί στο τοπικό επίπεδο. Ευχαριστούμε. Κύριο Ζωρολό. Ευχαριστώ. Σαν συμπέρασμα αλλά και αντιδρώντας τις παρεμβάσεις σας μιλήσατε για τον ανταγωνισμό. Ποια θα ήταν η καλύτερη χώρα όσον αφορά την ποιότητα ζωή στην εργασία. Μάλιστα, α κάνουμε ένα τέτοιο ανταγωνισμό μεταξύ μα, ας ανταλλάξουμε τι καλύτερε πρακτικέ, ας τι μεταφέρουμε μεταξύ μα, ας τι εφαρμόσουμε για να το πετύχουμε. Τώρα κάτι που τίθεται και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους πολιτικούς και τις κοινωνίες. Παλιά στις κοινωνίες μας είχαμε μια διακυβέρνηση από πάνω προς τα κάτω, τώρα είναι πιο οριζόντια. Οπότε ο κόσμος και οι μισθωτοί και οι επικεφαλείς των επιχειρήσεων πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν. Πρέπει να οργανώσουμε τη συμμετοχή αυτή. Είναι θέμα management, αλλά είναι και θέμα δημοκρατία. Επανερχόμεθα στο θέμα τη κοινωνική και οικονομική δημοκρατία και πώ την αντιλαμβανόμαστε στο σημερινό κόσμο. Όσο πιο κοντά είμαστε στην πραγματικότητα, τόσο πιο ρεαλιστές θα μπορούμε να είμαστε και τόσο καλύτερα θα μπορέσουμε να δώσουμε τις καλές λύσεις. Ανακλάδο, ανατομέα. Ο ρόλος του πολιτικού είναι να θέσει το πλαίσιο. Το πλαίσιο το οποίο θα οδηγήσει στη συνέχεια σε τέτοιου είδους εφαρμογές. Πρέπει επίσης κάποιες επιχειρήσεις να τις κοιτάξουμε ιδιαίτερα, επειδή είναι ιδιαίτερες από μόνες τους και αυτές είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν διαφορετικά. Δεν λέω ότι πρέπει να έχουμε χαμηλότερου στόχου και προσδοκίε όχι, αλλά πρέπει να υπάρχει συνοχή με την πραγματικότητα που ζουν οι επιχειρήσεις αυτές. Ο κοινωνικό διάλογο τώρα. Οι κοινωνικοί εταίροι φυσικά πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να τον υλοποιήσουν. Αλλά και η πολιτική παίζει ρόλο και γι' αυτό στρέφομαι και στην Επιτροπή. Φυσικά ο καθένα έχει διαφορετικού κοινωνικού διαλόγου στη χώρα του. Στο Βέλγιο τον έζησα, ήμουν, γενικό γραμματέα μια συνδικαλιστική οργάνωση και την πλήρωσα ήταν μια μέθοδος όπως εκλέγουμε τον Πάπα περίπου. Δηλαδή κλείνουμε τους ε, συνδικαλιστές στην εργοδοσία σε μια αίθουσα και τους λέμε «Να, αυτό είναι το θέμα, φροντίστε να συμφωνήσετε». Αν δεν συμφωνήσετε θα πάρουμε εμεί μια απόφαση που δεν θα σας αρέσει ούτε σε εσά τους συνδικαλιστές ούτε σε εσά την εργοδοσία. Βέβαια μερικές φορές λειτουργήσε καλά. Και αν θυμάμαι καλά την ιστορία, είναι όπως έγινε και στο Βαλντουσές, έτσι, με τις συμφωνίες ΣΕΣ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Περίνσκι. Ένα από τα ερωτήματα ήταν πώς μπορεί αυτό, αυτή η έρευνα να μετουσιωθεί σε πράξη. Και πιστεύω ότι ένα από τα στοιχεία είναι να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στις μεγάλες διαφορές αυτές οι οποίες ε, κυμαίνονται πολύ πάνω, πολύ κάτω από το μεσόωρο, είτε είναι διαφορές ε, τομεακές, είτε διαφορετικές γεωγραφικές κτλ. Διότι γνωρίζουμε ότι στους διάφορους κλάδους ε, της εργασίας οι διαφορές είναι έντονες και άρα απαιτούν διαφορετικές πρακτικές. Θα ήθελα να επανέλθω όμως και στο σχόλιο που έκανε ο κ. Σερβός προηγουμένως σχετικά με τις ε, νοσοκόμες οι οποίες έχουν σπουδάσει στην Ισπανία και όμως εργάζονται στην ε, Γαλλία. Ε, και στην Βουλγαρία έχουμε το ίδιο πράγμα. Εμείς έχουμε υψηλού επίπεδου εκπαίδευση και οι νέοι μας όμως αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο των σπουδών φεύγουν διότι βλέπουν, βρίσκουν πολύ ελκυστικές θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Επομένως χρειάζεται μεγαλύτερη γεωγραφική συνοχή, ε, χρειάζεται μία επανεκκίνηση της ε, βιομηχανίας. Το παράδειγμα της Κατερπιλάρα δείχνει ας πούμε την ανάγκη αυτή ακόμα περισσότερο. Και έγινε λόγος και για τις συνθήκες. Ας δούμε λίγο το άρθρο 3 της ε, συνθήκης, το οποίο ρητά αναφέρει την μέγιστη ανάγκη ε, ε, συνοχής σε όλα τα επίπεδα. Κατά αυτή την έννοια, η εταιρική σχέση, ιδίως η ε, κοινωνική εταιρική σχέση, είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ζήτημα λοιπόν είναι εάν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αυτές οι οποίες θα ε, λειτουργήσουν θετικά ε, έτσι ώστε και οι εργαζόμενοι να επιλέγουν ε, την θέση εργασίας τους με ικανοποίηση. Ξέρουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει αποδυναμωθεί, έχει όλο και λιγότερους όλο και λιγότερα μέλη και αυτό νομίζω πως οδηγεί σε αρνητικά συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Φόλτεν. Πρώτον, να σας πω ότι ήδη από σήμερα στην ε, ε, ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε την ε, έκθεση. Αλλά το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλα αυτά, όλες οι εξελίξεις Κοιτάξτε, ακούσαμε ε, και την ε, φιλανδική εμπειρία. Ε, νομίζω ότι ότι μπορούμε και να προωθήσουμε αυτή την εργασία, να ευαγγελίσουμε αυτόν τον καλό λόγο έτσι ώστε να υπάρξει μια ανταλλαγή πρακτικών. Νομίζω ότι πλέον είναι σαφές ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ε, προχωρήσουν στο σωστό δρόμο και επομένως μόνο κερδισμένοι όλοι μπορούμε να βγούμε από αυτή την κατέσταση. Ε, πάντως είναι πάρα πολύ θετικό που είχαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την εργασία σήμερα τώρα όσον αφορά κάποιες ερωτήσεις που ακούστηκαν. συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Είμαι βεβαία ότι θα υπάρξουν δυνατότητες ε, για περαιτέρω συζητήσεις και ώστε να απαντηθούν και ε, ερωτήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα απαντηθεί. Λοιπόν, τώρα σας καλώ όλους ε, σε γεύμα το οποίο θα δοθεί εδώ έξω. Θα ξεκινήσει τώρα και εμείς θα ξαναρχίσουμε την απογευματινή μας και δεύτερη συνεδρία στις μισή 14 και 30. Εδώ σε αυτή την ίδια αίθουσα, 2Q2. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή η συνεδρία γιατί αυτή η, ε, ο συνδυασμός ε, της ε, επαγγελματική ζωής και της υπόλοιπης ζωής είναι κάτι συναρπαστικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ακριβώς και αυτός είναι και ο, ο ο τίτλος της έρευνας υπάρχει ακόμα ε, περιθώριο διερεύνησης των δύο στοιχείων έτσι ώστε καλύτερα να συνδυαστούν μεταξύ τους. Λοιπόν, ε, σας καλώ ε, επομένως στο γεύμα εδώ έξω και θα ξαναρχίσουμε στις 2.30. Σας ευχαριστώ βέβαια και για την συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα.